Παρακαλώ τους κυρίους φωτογράφους και εικονολήπτας να εξέλθουν τις αιθούσεις διότι άρχεται η συνεδρία. Παρακαλώ, βγείτε. Nous puissions commencer nos travaux. Merci. Bon après-midi, Καλό σας απόγευμα, αγαπητοί συνάδελφοι και κυρία Γέλεβα και καλωσορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλοι γνωρίζουμε το στόχο της ακρόασης αυτής, που είναι ακριβώς η ακρόαση της κυρίας Γέλεβα, για να δούμε κατά πόσο έχει τα προσόντα και τις ικανότητες να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της Διεθνούς Συνεργασίας Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείριση Κρίσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χαρτοφυλάκιο που της επεφύλαξε ο πρόεδρος κ. Μπαρόσο. στις κατευθυντήριες γραμμές, λαμβάνοντας υπόψη το παράρτημα 17 του κανονισμού, εμείς ε, αξιολογούμε βάσει των ικανοτήτων τους επιτρόπους της ευρωπαϊκής Προσύλλευσης και της ε, προσωπικής τους ανεξαρτησίας. Ε, επίσης, εξετάζουμε τη δυνατότητα επικοινωνίας που έχουν. Θυμίζω επίσης ότι η υποψήφια επίτροπος πριν από την ακρόαση απάντησε γραπτός στο προπαρασκευαστικό ερωτηματολόγια. Σας έχουν διανεμηθεί δε οι γραπτές απαντήσεις. Πριν αρχίσουμε τα προφορικά, θα ήθελα να σας θυμίσω πώς θα διεξαχθεί η ακρόαση. Πρώτον, σύντομη δήλωση των πολιτικών ομάδων για τις προτεραιότητες στην ανθρωπιστική βοήθεια και τη διαχείριση των κρίσεων. Στη συνέχεια, η υποψήφια επιτροπός θα κληθεί να κάνει εισαγωγική δήλωση, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 λεπτά. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν 2 ώρες και 45 περίπου ερωτήσεων με ένα γύρο τραπέζις από κάθε πολιτική ομάδα, Ένα εκπρόσωπος. Σύμφωνα με την αρχή, ε, τη λεγόμενη του πινκ-πονγκ. 3,5 λεπτά το πολύ έκαστος και 45 δεύτερα για την ερώτηση, ένα λεπτό και 45 για την απάντηση, 30 δεύτερα για συμπληρωματική ερώτηση και 30 δεύτερα για συμπληρωματική και τελική απάντηση. 45 λεπτά ε, είναι ο ανώτατος χρόνος που αναλογεί σε κάθε βουλευτή και όσο πιο σύντομοι είσαστε τόσο πιο εύκολα θα απαντήσει η Επίτροπος και θα υπάρξουν και συμπληρωματικές ερωτήσεις και η συμπληρωματική εκάστοτε ερώτηση θα πρέπει να συνδέεται με την απάντηση της υποψηφίας Επιτρόπου και δεν θα πρέπει να αναφέρεται σε άλλα άσχετα θέματα. Και ως Πρόεδρος δεν ε, ε, διατηρώ το δικαίωμά μου να μην δεχτώ ερωτήσεις που θα είναι άσχετες. Έχουμε και σύντομη διαδικασία Catch the Eye, όποιον δει πρόεδρο, για θέματα που συμφώνησαν οι συντονιστέ και συνιστούν προτεραιότητε για την Επιτροπή μα. Οι βουλευτέ που επιθυμούν να λάβουν το λόγο στη διαδικασία αυτή θα έχουν 15 με 20 δεύτερα για να κάνουν την ερώτησή του. Και παρακαλώ την Επίτροπο να πει πάρα πολύ σύντομε απαντήσει τη. Σα ενημερώνω ότι για το χρόνο αγόρευση, θα δοθεί προτεραιότητα στα τακτικά μέλη και στα πνευματικά μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης. Επίσης προβλέψαμε λίγο χρόνο που θα καλέσω την υποψήφια Επίτροπο να συγκεκριμενοποιεί την απάντησή της ή να ε, απαντά με τρόπο πλήρη να τις συμπληρώνει εφόσον το ζητούν οι πολιτικές ομάδες. Ε, είχαμε καλέσει και την Επιτροπή Περιβάλλοντος και την Επιτροπή Εξωτερικών να συμμετέχουν στη ε, ακρόαση αυτή. Στο τέλος της ακρόασης θα καλήσω την κυρία Γέλεβα να κάνει μια σύντομη καταληκτική δήλωση εάν το επιθυμεί. Έχουμε διερμηνία σε όλες τις γλώσσες. Όλοι οι ομιλητές μπορούν λοιπόν να ε, ομιλούν τη μητρική τους. Παρακαλείστε όμως να λαμβάνετε υπόψη ε, την ανάγκη διερμηνίας και να μην μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα. Και ε, στο web streaming ε, μεταδίδεται απευθείας στο διαδίκτυο η συνεδρίαση και βιντεοσκοπείται και θα παραμείνει στην ίδια ιστοσελίδα. Επιπλέον θα έχουμε πλήρη πρακτικά, αναλυτικά, γραπτά το συντομότερο. Αφού σας είπα όλα αυτά, προχωρούμε στην ακρόασή μας και αρχίζουμε από τις δηλώσεις των πολιτικών ομάδων. E. Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα το λόγο ο κύριος Φίλιπ Κασμαρέκ για να κάνει την αρχική δήλωση της ομάδας. Ε, Ευχαριστώ. Θα μιλήσω πολωνικά γι' αυτό. Βάλτε τα ακουστικά σας παρακαλώ. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η συνθήκη της Λισαβόνας αναφέρει την ανθρωπιστική βοήθεια για πρώτη φορά σαν μία από τις εξωτερικές πολιτικές. Και για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουμε μία επίτροπο, έναν επίτροπο που θα είναι υπεύθυνο για την ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει την ανθρωπιστική βοήθεια με πολύ σοβαρό τρόπο. Και ότι θέλει να ενδυναμώσει το ρόλο που παίζει σε αυτόν τον τομέα. Νομίζω ότι είναι ένα καλό βήμα, ένα σωστό βήμα και είμαστε ικανοποιημένοι που υπάρχει ένας τέτοιος ε, επίτροπος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθήσει τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή των δράσεών της. Επίσης θα πρέπει να είναι έτοιμη για να αντιμετωπίσει όλο και μεγαλύτερες δυσκολίες, όλο και μεγαλύτερες προκλήσεις και αυτό το είδαμε και πέρυσι. Μία από αυτές τις προκλήσεις είναι η ουδέτερη και αποτελεσματική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας η πραγματικότητα δεν είναι λόγος για αισιοδοξία. Ο κύριος Μπέρμαν. Ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα τεράστιο οργανωτικό πρόβλημα. Ε, διαιρούνται τα χαρτοφυλάκια σε πολλούς επιτρόπους. Τα μέσα αναπτυξιακής βοήθειας ε, είναι της Lady Ashton. Ο κ. Πίμπαλξ ασχολείται με τη EuroPaid και εσείς ε, με τα ψυχία μεταξύ των οποίων και η ανθρωπιστική βοήθεια. Υποτίθεται ότι η δράση αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι τρεις ε, επίτροποι. Αυτό είναι συνταγή για συγκρούσεις και έλλειψη συνοχής. Αντί να υπάρχει ένας έντονος ρόλος για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για τη μείωση της στόχη, ο κ. Μπαρόσο θέλει να διαιρέσει τις εξουσίες. Ε, η ανθρωπιστική βοήθεια, η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια θα έπρεπε να είναι αρμοδιότητε ενό επιτρόπου και να είναι υπεύθυνο για όλα αυτά τα θέματα. Αλλά δυστυχώ ο Μπαρόζο το αγνοεί αυτό. Δεν ε, περιμένω εσεί να ξεκαθαρίσετε αυτό το χαμό που γίνεται. Αλλά πώ θα εξασφαλίσετε ότι η χρηματοδότηση τη ανθρωπιστική βοήθεια δεν, θα ε, δεν θα γίνει με τρόπον αποτελεσματικό. Πώ θα προχωρήσετε ε, πώς θα εξασφαλίσετε το στενό στόχο της, ε, και τη συμπληρωματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας με τις διάφορες εξελίξεις. Πριν να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, κυρία Γέλεβα, θα ήθελα να μας εξηγήσετε γιατί αντίθετα από τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως ε, βουλευτής δεν αναφέρατε στη δήλωση συμφερόντων το 2008 και το 2009 ότι είσαστε μάνατζερ της δικής σας εταιρείας consulting. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Γκέρεντς από τους φιλελευθέρους. Ευχαριστώ. Τα καθήκοντα της μελλοντική Επιτρόπου για την ανθρωπιστική δηλαδή βοήθεια είναι βαριά και δυσβάστακτα. Αλλά και σημαντικά διότι πρέπει να δώσει μια απάντηση σε δύσκολες καταστάσεις και μάλιστα γρήγορα και χωρίς μεροληψία. Αυτό είναι προφανές αλλά σημαίνει απ' την άλλη ότι εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και στρατιωτικές και ανθρωπιστικές δικαιοδοσίες δεν πρέπει να βλάπτουν η μία την άλλη και ιδίω η ανθρωπιστική βοήθεια να εμποδίζεται από τις στρατιωτικές δραστηριότητες. Ε, Ως ανταπόκριση σε αποτυχία βέβαια πρέπει να αναλάβετε τα καθήκοντά σας. Γιατί, διότι πρέπει να αναλάβετε δραστηριότητες αναπτυξιακές και διορθωτικές των καταστάσεων. Άρα να συνεργάζεστε με όλους και θα ήθελα να μου πείτε ποιες δυνατότητες και ποια όρια βλέπετε στη δραστηριότητά σας ως έχει αυτή τη στιγμή η Κομισιόν. Πώς η κυρία Κέλλερ των Πρασίνων. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να τονίσω μερικά σημαντικά σημεία για μας τους Πρασίνους. Μεγάλο τμήμα των καταστροφών που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσετε είναι δομικά προβλήματα για τα οποία εν μέρη υπεύθυνη είναι και η Ένωση. Πρέπει λοιπόν να θυμάστε και εσείς και ολόκληρη η Ένωση αυτούς τους δομικούς λόγους που δημιουργούν τέτοιες δύσκολες καταστάσεις και καταστροφές. Παραδείγματος χάρη τις κλιματολογικές αλλαγές. Ανησυχούμε διότι όλο και γίνονται λιγότεροι οι διαχωρισμοί που υπάρχουν μεταξύ θεμάτων ασφαλείας και θεμάτων ανθρωπιστικών και άλλων. Η Βουλγαρία, η χώρα σας, δεν έχει ακόμη μία, καμία σαφή στρατηγική αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων και είναι ίσως η μόνη χώρα που δεν το έχει κάνει. Και παρόλα αυτά θα ήθελα να μας πείτε πώς θα μπορέσετε να αναλάβετε αναπτυξιακά θέματα αφού η Βουλγαρία δεν κάνει τίποτα. Τέλος, σε μία συνέντευξη με τους Financial Times στη Γερμανία υπήρχαν ορισμένα χάσματα ή λάθη στις δηλώσεις συμφερόντων που είχατε κάνει. Δεν θα μπορούσατε να είχατε υπάρξει λίγο πιο διαφανής. Ο κύριος Σαντήλ της Ουσλαέρ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Εμείς έχουμε τρία σημεία να θίξουμε. Πρώτον, η προετοιμασία και διαχείριση κρίσεων. Πρέπει να βρούμε κάποιον τρόπο να μαζέψουμε κάπου στρατηγικά αποθέματα. Και δική σας ευθύνη θα είναι αυτό. Δεύτερον, Δεύτερον, πρέπει να προετοιμαζόμαστε και για τις διατροφικές κρίσεις που φαίνεται ότι ετοιμάζονται στην Αιθιοπία και αλλού και χρειάζονται και εκεί αποθήκες. Άρα περισσότερα, μεγαλύτερα κονδύλια από όσα διαθέτουμε. Και αυτό δική σας δικαιοδοσία. Και τρίτον, να βασιστούμε σε με ορισμένες μήκη οργανώσεις οποίες, για τις οποίες ενδιαφέρομαι και εγώ πολύ. Δυστυχώς δεν είναι όλες οι ανθρωπιστικές οργανώσεις ίσες, μερικές έχουν ε, πολύ αρνητική δράση και θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να διαφοροποιήσουμε τις ε, καταλληλότερες από τις ακαταλληλότερες. Εκείνε δηλαδή που δαπανούν 75 με 80% του προπολογισμού τους μόνο για τα λειτουργικά τους έξοδα, άρα δεν κάνουν στην ουσία τίποτα. Και αυτό δική σα δικαιοδοσία θα είναι. Θα τα ξαναθίξω με ερωτήσει, αλλά αργότερα αυτά τα τρία σημεία. Η κυρία Σινμεαρ τη Γκουε. Ευχαριστώ. Κυρία Γέλεβα, ορίζουμε τη συνένωση της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ε, αντιμετώπισης των κρίσεων και είμαστε υπέρ ε, της πιο ενεργού συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το τομέα. δική μας η αριστερή ομάδα ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την άποψή σας για το πώς θα οργανώσετε τη συλλογή και οικονομικών πόρων και πώς θα το επιβάλλετε αυτό, γιατί μέχρι τώρα έχουμε ε, ασαφείς και γενικές και αόριστες υποσχέσεις των κρατών μερών, αλλά όταν έρθει η ώρα να βάλουν το χέρι στην τσέπη, τα κράτη-μέλη εμφανίζουν απροθυμία. Επίσης, τι γίνεται με την πρόληψη των κρίσεων. Είναι στοιχείο του δικού σας χαρτοφυλακίου αυτό και σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, τι γίνεται με τις φτωχές αναπτυσσόμενες χώρες. Θα τις υποστηρίξουμε ε, συγκεκριμένα και σε ποιο βαθμό θα φροντίσετε τα αντίστοιχα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να συμμετέχει όσο μπορεί με τις δυνατότητές της ενεργά έτσι ώστε η ανθρωπιστική βοήθεια, κυρίως η πρόληψη των κρίσεων ε, και η αντιμετώπιση των κρίσεων είναι κάτι το οποίο να μας απασχολεί. Υπάρχει μια διευκόλυνση μετά το τσουνάμι ενός δισεκατομμυρίου αλλά αυτό δεν ε, αξιοποιήθηκε επαρκώς. Η Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια. Je donne la parole à Madame Sinclair de EFT pour une minute. Για 1,5 λεπτό, η κυρία Σενκλέρα από την ε, Ευρώπη για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία. Madame Sinclair n'est pas là. Σιάζει κυρία Σανκλέρ. Ε, τότε θα δώσω το λόγο στην κυρία Γέλεβα για να κάνει την εισαγωγική της δήλωση, την πολιτική. για 10 λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, κύριε μόνιμα, ε, ε, εισηγητά, κυρία, συγγνώμη, αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη τιμή για μένα, ευκαιρία που έχω να παρευρίσκομαι ως υποψήφια επίτροπος. Με τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Σαββόνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Αυτό διανοίγει μια τεράστια δυνατότητα και ευκαιρία για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να φέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της και να ενισχύσουν το ρόλο της Ευρώπης παγκοσμίω ανέκαθεν εργαζόμουν για μια Ευρώπη ισχυρή και ενωμένη που να υπερασπίζεται τις αξίες της όπως είναι η αξιοπρέπεια, η ελεγγύη και θεωρώ προνόμιο το γεγονός ότι ε, ευθύνη μου θα είναι να εκπροσωπώ την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και τις αξίες της ε, και εντός και εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων. Εξελέγην δις ευρωβουλευτής και γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διάλογο με το κοινοβούλιο σας. Το κοινοβούλιο ανέκαθεν ήταν αποτελεσματικό, ταχύ και υποστηρικτικό ε, στο ρόλο του. Είμαι δεσμευμένη προς την κατεύθυνση αυτή να συνεχίσουμε και να ενισχύσουμε την καρποφόρο αυτή συνεργασία ε, βασιζόμενη στις ισχυρές βάσεις των προκατόχων μου Έμπο Μονίνο, Πάουλ Νίλσον, Λουίς Μισελ, ε, Κάρλ Ντεχόχτ και Σταύρου Δήμα. Η συνεργασία αυτή θα είναι ουσιαστική διότι αντιμετωπίζουμε διπλή πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και της οικονομικής κρίσης. Οι σειράξεις και οι θεομηνίες δεν σέβονται σύνορα. Σήμερα έχουμε 42 εκατομμύρια εκτοπισμένους παγκοσμίως ο αριθμός των θεομηνιών που συνδέονται με τις κλιματικές αλλαγές έχουν τριπλασιαστεί το τελευταίο διάστημα, τελευταία δεκαετία. Στην Ευρώπη οι φυσικές καταστροφές καταλήγουν σε μια τεράστια λίστα ανθρωπίνων εγωδιών και κοστίζουν στον Ευρωπαίο φορολογούμενο 15 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, συχνά οι πιο ευάλωτοι, οι γυναίκες, τα παιδιά και οι φτωχοί είναι εκείνοι που πλήγονται πιο σκληρά. Εν ώψη αυτού του δραματικού σενάριου, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να οικοδομήσει μια ισχυρή δυνατότητα αντιμετώπισης των κρίσεων. Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ε, και να αξιοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα τους ε, διαθέσιμους πόρους. Γι' αυτό ο ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής μου θα είναι ο συντονισμός. Το μελλοντικό μου χάρτοφυλάκιο ε, συγκεντρώνει μια ισχυρή διεθνή παρουσία και ε, την πραγματογνωμοσύνη και τους πόρους της Κομισιόν και ε, των κρατών μελών στους τομείς της ανθρωπιστικής βοήθειας και της πολιτικής προστασίας όπως ε, αναφέρεται στην έκθεση Μπαρνιέ του 2006 αντιπροσωπεύει μια εντυπωσιακή βάση για ε, μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της Ένωσης σε αντιμετώπιση κρίσεων σε επίγουσες περιπτώσεις. Αυτό που θέλουμε είναι μια ταχεία και σωστή ανταπόκριση σε οποιοδήποτε είδους κρίσες. Στο διεθνή χώρο θα συνεργαστώ με ε, ευρεία κλίμακα οργανώσεων μεταξύ αυτών ε, τον ΟΗΕ, το παγκόσμιο πρόγραμμα ε, επιστημιστικό, ε, την ύπατη αρμοστία για τους πρόσφυγες, τη UNICEF και μια σειρά ε, περιφερειακών και τοπικών οργανώσεων. Στα γερμανικά τώρα. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, η ανθρωπιστική βοήθεια δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα μιας καλής πολιτικής. Εγώ θέλω να βασιστώ να οικοδομήσω πάνω σε αυτή τη βάση και δεν θα διστάσω να στείλω σαφή μηνύματα και σε πρωτεύουσε και σε περιοχές που γνωρίζουν κρίση. Εδώ προσβλέπω και σε στενή συνεργασία με την ύπατη εκπρόσωπο και αντιπρόεδρο κυρία Άστον. Επίσης θα ήθελα να σας παρουσιάσω, μου επιτρέπετε, ε, κάποιες προτεραιότητές μου. Θα φροντίσω να ενισχυθεί ε, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Αυτό που με ενδιαφέρει εδώ είναι να αντιμετωπιστούν βίες ε, και ομές ε, μέθοδοι πολέμου, βία σε γυναίκες και παιδιά ως πολεμικά μέσα. Επιπλέον θα ασχοληθώ ε, ιδιαίτερα με τους ανθρώπους που βρίσκονται ε, σε κρίσεις και ε, αντιμετωπίζουν πολλά δεινά. Δεν αρκούν μόνο τα χρήματα. Θα πρέπει να μπορούν και οι διάφοροι ανθρωπιστικοί φορείς να εργάζονται επί τόπου. Και το τελευταίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και απαραίτητο, γιατί πολύ συχνά οι κυβερνήσεις αρνούνται την ίδια την ύπαρξη τέτοιων κρίσεων ορισμένε κυβερνήσεις εντός των συνόρων τους αρνούνται καν το γεγονό ότι υπάρχει μια ανθρωπιστική κατάσταση ε, επίγουσα. Νταρφούρ, Σρι Λάνκα, Ερυθρέα, θυμίζω απλά και μόνο ορισμένε περιπτώσει. Άλλη προτεραιότητα είναι σαφής διαχωρισμός ε, στρατιωτικών δραστηριοτήτων και ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων. Όλο και πιο συχνά ε, στρατιωτικές ε, και τακτικές φιλοδοξούν στο να κερδίσουν τις καρδιές των ανθρώπων. Όλο και περισσότερο υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Και πολύ συχνά ε, οι ε, δράστες της ανθρωπιστικής βοήθειας, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις γίνονται στόχος. Και εγώ θα ήθελα να βελτιώσω ε, την ασφάλεια. Επί το 2008 θανατώθηκαν 122 υπάλληλοι ανθρωπιστικών οργανώσεων. Περισσότεροι από ωκεανόκρανους. Γι' αυτό προσωπικά θέλω εδώ και τώρα να αποτίσω ένα φόρο τιμή στους ανθρώπους αυτούς για ε, τον επαγγελματισμό τους και ε, που πλήρωσαν με το υψηλότερο τμήμα με τη ζωή τους. Αφγανιστάν, Γάζα, Σρι Λάνκα, Νταρφούρ, Σομαλία, Τσάντ, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Σας αναφέρω μερικά παραδείγματα μόνο. Όλα αυτά είναι παραδείγματα πάρα πολύ καλά γνωστά ε, για τα προβλήματα που σας ανέφερα. Το να αντιμετωπίσουμε αυτά τα περίπλοκα προβλήματα θα είναι μία από τις βασικές μου αρμοδιότητες. Και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις προτάσεις σας. Ελπίζουμε να έχουμε και ένα καλύτερο μέλλον. Μόλις έχει περάσει η πιο σοβαρή ε, φάση μιας κρίσης χρειάζεται οικοδόμηση του μέλλοντος. Γι' αυτό ε, θα πρέπει να γίνει μια σωστή μετάβαση από την ανθρωπιστική βοήθεια, από τη βοήθεια προς την ελπίδα. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν θα αποτελέσει προτεραιότητα για μένα και το έργο μου να έχουμε μια συνεκτική και καλά συντονισμένη ευρωπαϊκή παρουσία. Εδώ θα συνεργαστώ στενά με τη Βαρόνη Άστον και τον Επίτροπο κύριο Πίλμπαρξ. Στα βουλγαρικά τώρα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σε ό,τι αφορά ε, την πολιτική προστασία Πρέπει να σας πω ότι εδώ θεωρώ ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία στην ευρωπαϊκή διάσταση. Καλύτερη προετοιμασία, καλύτερο συντονισμός. Το ε, κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την πολιτική του προστασία. Αν έχουμε πληροφορίες για τον αριθμό των ε, νοσοκομείων, των υλικών, των τεντών που έχει κάθε κράτος μέλος ε, και αν ξέρουμε πού ακριβώς χρειάζονται θα μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να αλληλοβοηθηθούμε πιο αποτελεσματικά. Νομίζω ότι αυτή είναι η σημασία της νέας ρήτρα αλληλεγγύης. Νομίζω ότι εκεί ε, εδράζεται το ευρωπαϊκό πνεύμα. Επομένως, με στενή συνεργασία ε, με την Επίτροπο Μάλστρομ θα εξυγχρονίσω τον ε, μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης και θα εμπλέξω όλους τους ενδιαφερόμενους. Θα έχουμε ένα αρχηγείο και ένα επιχειρησιακό κέντρο ικανό να συντονίσει τη βοήθεια σε περίπτωση κρίσης, προκειμένου να βοηθήσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες και τους υπόλοιπους κληθισμούς ε, που κατοικούν εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή θα είναι μια συνολική προσέγγιση που θα καλύπτει όλες τις φάσεις από την πρόληψη μέχρι την αποκατάσταση. Και τέλος, μετά από ευρείες διαβουλεύσεις θα παρουσιάσω και μία πρόταση για την εφαρμογή και τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών ε, με βάση τα όσα επιτάσσει και η συνθήκη της Λισαβόνας. Αξιο τη μαμέλη αυτή της, ξέρω, μαμέλη του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, γιατί το Κοινοβούλιο ήταν πάντα παρόν. Ε, τονίσατε πάντα τη σημασία του, ενός κατάλληλου προϋπολογισμού για την ανθρωπιστική βοήθεια που θα συμπεριλαμβάνει και την προετοιμασία έναντι των καταστροφών και ζητήσατε από την Κομισιόν να έχει ισχυρότερες δομές και δυναμικό στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Οι πολιτικές μου προτεραιότητες ε, σχεδιάζονται για να αντιμετωπίσουν πιστούν ακριβώς τα αιτήματά σε αυτόν τον τομέα και θεωρώ ότι αυτή η ακρόαση είναι το πρώτο βήμα για να υπάρξει μια ε, εποφελή συνεργασία. Περιμένω με ανυπομονησία να συνεργαστούμε και με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια κοινή προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε ότι αυτό το νέο χαρτοφυλάκιο δημιουργεί και μεταφράζεται σε πραγματικά και αυτά αποτελέσματα. Η βοήθεια που θα δώσουμε ε, δεν είναι απλώς υλικό ε, και υλική βοήθεια. Είναι ελπίδα. Ελπίδα για ένα καλύτερο και πιο ασφαλές ε, και πιο λαμπρό μέλλον. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Τώρα θα έχουμε μία ε, διαδικασία Catch the Eye για πέντε λεπτά για το πρόβλημα του ε, λύματος ε, στο, στη δημοκρατική, στο ανθρωπιστική βοήθεια. Για τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν ανάμεσα στην αποκατάσταση, την επίγουσα βοήθεια και την ανάπτυξη. Και το συντονισμό που θα πρέπει να εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Γκερέρο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να παρακαλέσω την υποψήφια να αναπτύξει λίγο περισσότερο τη γενική της αντίληψη για τα προγράμματα αποκατάστασης. Για τη μετάβαση ακριβώς από την άμεση αντιμετώπιση των κρίσεων την επίγουσα. δεύτερο λεπτά, ε, δευτερόλεπτα η ερώτηση λέει η πρόεδρος. Έχετε το λόγο. regionale și Πώς ε, αντιλαμβάνεστε τη συνεργασία με τους ε, διάφορους περιφερειακούς οργανισμούς και με τον ΟΗΕ σε περίπτωση κατεπήγοντων ε, προβλημάτων, φυσικών καταστροφών κτλ. Ο κύριος Στένσον έχει το λόγο. Υπάρχουν ομάδες, οι πρόσφυγες ας πούμε και η Ρώμα, που συχνά χαρακτηρίζονται παράνομοι πληθυσμοί που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Συχνά μιλάμε για την ανθρωπιστική βοήθεια εκτό των συνόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώ μπορείτε να δώσετε βοήθεια για αυτού του ανθρώπου που τη χρειάζονται πραγματικά. Ο κύριο Λάμστορφ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ως Πρόεδρος ομάδα εργασία για τι σχέσει με ε, τον ΟΗΕ, σα ρωτώ πώ. Ε, φαντάζεστε συγκεκριμένα τη συνεργασία με την ύπατη αρμοστία για τους ε, πρόσφυγες και ιδιαίτερα με τη UNICEF για τα παιδιά που ζουν σε τέτοιες ε, καταστάσεις κρίσης. Ο κύριος Φίσα Σαγιάλα. Τελευταία ερώτηση με το ΚΑΤΣΙΑ. Ευχαριστώ. Ποια διαφορά βλέπετε ανάμεσα στη διεθνή συνεργασία που είναι δικό σας θέμα και την αναπτυξιακή βοήθεια που είναι στο χαρτοφυλάκιο του κυρίου Πίβαλξ. Έχετε το λόγο για τρία λεπτά, κυρία Γέλεβα. Ευχαριστώ. Καταρχήν, θα ήθελα να πω ότι κενά στην ανθρωπιστική βοήθεια υπάρχουν και είναι σοβαρό το θέμα. Και εγώ θα ήθελα να το αντιμετωπίσω στα πλαίσια του νέου χαρτοφυλακίου μου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα λόγω του καταμερισμού των εξουσιών μεταξύ της αναπτυξιακής βοήθειας και της ανθρωπιστικής βοήθειας. Δεν υπάρχει πρόβλημα αυτά τα δύο χαρτοφυλάκια. Στο παρελθόν ε, είχαμε κάποιες πρακτικές συνεργασίας πολύ καλές για χώρε που δεν ανήκαν στην ομάδα ΑΚΕ και εκεί είχαμε μοιρασμένα αυτά τα χαρτοφυλάκια. Θα ήθελα τώρα να απαντήσω τις πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις σας, πολύ συγκεκριμένα. Για τα προγράμματα αποκατάστασης. Θα ξέρετε ίσως ότι στο χαρτοφυλάκιό μου έχουμε ένα προϋπολογισμό για την ανθρωπιστική βοήθεια Έχουμε τον τρίτο πυλώνα που είναι ε, η πρόληψη από τις φυσικές καταστροφές. Θέλουμε να υπάρξει στενότερη σχέση μεταξύ αποκατάστασης και αναπτυξιακής βοήθειας. Φυσικά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει διαφορετική φύση σε αυτές τις δύο πολιτικές, της ε, αναπτυξιακής ε, πολιτικής και της ε, ανθρωπιστικής βοήθειας. Η ανθρωπιστική βοήθεια έχει σαν σκοπό να σώσει τη ζωή των ανθρώπων και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Στην περίπτωση της αναπτυξιακής πολιτικής που συμπεριλαμβάνει και το θέμα της αποκατάστασης, θα πρέπει να μας υποστηρίξουν και οι κρατικοί φορείς στην εν χώρα. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία και θέλω να την ενδυναμώσω αυτή τη συνεργασία στις εκάστοτε χώρες με τις τοπικές αρχές, αλλά φυσικά μην ξεχνάμε και τα, τις αρμοδιότητες του συναδέλφου μου, του κ. Πίμπαλξ, ε, για τις περιφερειακές οργανώσεις τώρα και τον ΟΗΕ. Στα πλαίσια του χαρτοφυλακίου μου ε, υπάρχουν θετικές επιπτώσεις από τη διεθνή συνεργασία. Γιατί αυτό σημαίνει ότι θα συνεργαστούμε και με τον ΟΗΕ και τις οργανώσεις του ΟΗΕ, οι οποίες ε, δραστηριοποιούνται ε, επιτόπου και παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια με την OCHA και στην περίπτωση των και για τους πρόσφυγες και τους ε, εσωτερικά εκτοπισμένους θα συνεργαστούμε με την ύπατη αρμοστία προσφύγων. Σας παρακαλώ κυρία Γιάλεβα και εσείς να σέβεστε το χρόνο. Euh, και τώρα ακολουθεί ο πρώτος ε, γύρος ε, ερωταποκρίσεων. Σας θυμίζω τη διάφρωση. 45 δεύτερη ερώτηση, 1,5 λεπτό η απάντηση και συμπροματική ερώτηση 30 δευτερολέπτων με απάντηση επίσης 30 δευτερολέπτων. Α, έκανα λάθος. Ένα λεπτό και 45 δεύτερα η απάντηση. Τα έχουμε πολύ συγκεκριμένα ρυθμίσει. Ο κύριος Γκέι Μίτσελ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλησπέρα σας κυρία Γέλεβα. Δεν είναι μόνο λεφτά η υπόθεση του χαρτοφυλακίου σας, όπως είπατε και ίδια πολλά έχουν να κάνουν με τον προγραμματισμό, με την προετοιμασία και την πρόληψη των αναγκών. Με πρόβλεψη. Πώς λοιπόν θα κάνετε αυτό τον προγραμματισμό για να καταλάβουμε και πώς θα συνεργαστείτε μαζί μας στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή να μην περιμένουμε μόνο να αντιδρούμε αλλά να προλαμβάνουμε κιόλας ε, κρίσεις και περιβαλλοντικές ε, και αναπτυξιακές και θεομηνίες. Κυρία Γέβελα έχετε το λόγο. Θα είμαι πολύ συγκεκριμένη. Εγώ είμαι ανοιχτή στο διάλογο με το Κοινοβούλιο και συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να είμαστε δραστήριοι και όχι να αναμένουμε μόνο να συμβεί η κρίση, να μας συμβεί. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε μια άμεση απάντηση στην κρίση που να βασίζεται στην ανάλυση αξιολόγηση των αναγκών. Και με κοινωνική προστασία και με ανθρωπιστική βοήθεια μπορούμε να διασφαλίσουμε καλύτερο συντονισμό επιτόπου μεταξύ κέντρου και εμπειρογνωμόνων τουλάχιστον δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε μία πρώτη αξιολόγηση αναγκών για τις ε, περιοχές όπου σημειώνονται έκτακτες θεομηνίες ή καταστροφές. Δεν είναι μόνο τα χρήματα, αλλά χρειάζεται κυρίως μεγαλύτερη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Επόμενη ερώτηση. Ευχαριστώ. Από ό,τι είπε η υποψήφια επίτροπος φαντάζομαι ότι αυτά τα ενεργά σχέδια για την πρόληψη και όχι μόνο θεραπεία των κρίσεων θα αφορούν και την πρόληψη. Ναι, καλό είναι να υπάρχει η δυνατότητα ανάλυσης σεναρίων και πρόγνωσης και όχι μόνο αντίδραση σε κρίσεις που έχουν ήδη ξεσπάσει. Και αυτό είναι δυνατόν γιατί έχουμε πολύ καλούς επαγγελματίες στις υπηρεσίες μας. Η Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ έχει τη δυνατότητα να αναλύει εκ των προτέρων να κάνει αξιολογήσεις ή να αναλύει τις λεγόμενες ξεχασμένες κρίσεις. Και έτσι μπορεί να υπάρχει καλύτερο σχεδιασμός και προσχεδιασμός και καλύτερος σχεδιασμός με όλα τα μέσα που διαθέτουμε. Θα έλεγα λοιπόν ότι έχουμε πραγματικές δυνατότητες βελτίωσης καλύτερου συνδυασμού μεταξύ τεχνικών μέσων, ε, συνδυασμού όλων των μέσων που διαθέτουμε. Άρα χρειάζεται και η προετοιμασία σεναρίων εκ των προτέρων για θέματα ας πούμε κλιματολογικών αγωγών. Κάσιμαν. Ευχαριστώ. Κυρία Γέλεβα. Θα ξέρετε ότι ακούγονται φήμες και αντίφημες. Εμείς στην Επιτροπή μας ασχολούμαστε μόνο με γεγονότα. Γι' αυτό δεν θα ρωτήσω συμπληρωματική ερώτηση παρά μόνο το εξή. Στη δήλωση συμφερόντων που κάνατε, σύμφωνα με τη θεοντολογία για του επιτρόπου, υπάρχει τίποτε που παραλείψατε και που θα θέλατε τώρα να μα το πείτε για προηγούμενα συμφέροντα που δεν δηλώσατε. Μήπως, κυρία Γέλεβα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κάσμαρ για αυτήν την ερώτηση. Θα ήθελα να σας πω τον προτέρων ότι ποτέ δεν σχολιάζω φήμες που ακούγονται στον τύπο. Ιδίως για ό,τι ακούγεται για την προηγούμενη ζωή μου. Εδώ έχουμε έρθει να συζητήσουμε σημαντικά προβλήματα, ανθρωπιστική βοήθεια, αντιμετώπιση κρίσεων και τέτοια. Επομένως, και επίσης πώς να βοηθήσουμε, πώς να βοηθήσουμε ανθρώπους. Πώς να τους αποφύγουμε συμφορές. Αλλά εγώ δεν έχω τίποτα να κρύψω. και δεν υπάρχει τίποτα που να αρνηθώ να το απαντήσω ενώπιον της διακεκριμένης σας επιτροπής. Γι' αυτό δηλώνω ότι είμαι δημόσιον πρόσωπον από το 2007 και έχω δηλώσει ό,τι έπρεπε να δηλώσω. Μία φράση ακόμα. Όλες οι φήμες κατά του συζύγου μου ή εμού είναι τελείως αστήρικτες. Και τώρα ας παραμείνουμε στα θέματα που μας ενδιαφέρουν παρακαλώ. Συμπληρωματική όχι. Ο κύριος Γκέριντς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ερώτημά μου αφορά τη δυνατότητα ανταπόκρισης της Ένωσης σε καταστάσεις που απαιτούν την παρέμβαση της υπηρεσίας σας. Βασικά οι δυνατότητες αυτές προέρχονται από τα κράτη-μέλη βέβαια, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση καθεαυτήν δεν έχει τέτοιες δυνατότητες. Ερωτώ λοιπόν, οι δυνατότητες αυτές ανταπόκρισης, καταστάσεις κρίσεων, θεομηνιών, σειράξεων είναι επαρκής. Δηλαδή, Πώς θα αντιμετωπίζατε μια έλλειψη δυνατοτήτων σε αυτόν τον τομέα, πώς. Κυρία Γέλεβα. Ποτέ δεν είναι αρκετέ οι δυνατότητε για καμία κρίση. Αντιμετωπίζουμε δε ιδιαίτερα δύσκολου καιρού, όχι μόνο οικονομική κρίση και δημοσιονομική, αλλά και κλιματολογική. Κάτι και πρέπει να πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας την κατάσταση αυτή. Γι' αυτό θα ήθελα να σας απαντήσω ότι αφού υπάρχει κοινωνική προστασία και ανθρωπιστική βοήθεια για πρώτη φορά προβλέπετε θα διαβεβαιώνω ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να υπάρχει καλύτερη προετοιμασία μιας ανταπόκρισης, αλλά όχι μόνο ανταπόκρισης, αλλά και πρόληψης και εκπαίδευσης και άρα γενικά χρησιμοποίηση όλων των δυνατοτήτων που μου δίνει η θέση αυτή και θα ζητήσω από τα κράτη-μέλη να είναι και εκείνα πιο ενεργά ως προς την προετοιμασία αλλά και ως προς τη συμβολή που πρέπει να χορηγήσουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν στο πληρέστερο όλα τα μέσα που διαθέτουμε. Και έτσι να είμαστε προετοιμασμένοι. συμπληρωματική του κυρίου Γκέρεντ. Η συμπληρωματική αφορά την κατανομή των δικαιοδοσιών μεταξύ κρατών μελών. Θέλετε να ζητήσετε από τα κράτη-μέλη να κάνουν προσπάθειες σε συγκεκριμένους τομείς ώστε η προσπάθεια του ενός να αναλογεί κάπως την προσπάθεια του άλλου, ανάλογα βέβαια με το ΑΕΠ τους και τις δυνατότητές τους. κυρία Γελεβο, Η ανταπόκριση σε κρίσεις και θεομηνίες είναι η πρώτη φάση, σε πρώτη φάση εθνική. Έχουμε όμως τώρα τη δυνατότητα σύμφωνα με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης για καλύτερη προετοιμασία σε ενωσιακό επίπεδο και κινητοποίηση των δυνατοτήτων μας, ώστε να δείξουμε, να επιδείξουμε καλύτερα την αλληλεγγύη μας. Με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να τηρεί όλος ο κόσμος το χρόνο του. Η κυρία Ζαγκεντίνη. Ας το πω, ε, κυρία Γέλεβα, είπατε ότι είστε δημόσιον πρόσωπον. Τα δημόσια πρόσωπα δεν έχουν ιδιωτική δημοσιονομική ζωή, ούτε οι σύζυγοί τους. Έτσι λέει η δεοντολογία. Οι συνάδελφοι ζήτησαν, ρώτησαν πράγματα που δεν τα απαντήσατε. Θα ξαναρωτήσω λοιπόν. Γιατί δεν αναφέρατε τα συμφέροντά σας στο Global Consult το 2008 και 2009 την εποχή που το βουλγαρικό επιμελητήριο έδειχνε ότι είχατε τέτοια συμφέροντα ως ιδιοκτήτρια της εταιρείας. Γιατί. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι έχω δηλώσει ό,τι έπρεπε να δηλώσω. Ό,τι ήμουν υποχρεωμένη να δηλώσω. Και οι ειδικευμένε υπηρεσίες και οργανισμοί της Βουλγαρίας μου το έχουν επιβεβαιώσει. Έχω ετοιμάσει έναν τεράστιο φάκελο με επίσημα έγγραφα και στα βουλγαρικά και στα αγγλικά. Διότι ανέμενα αυτή την ερώτηση, την ανέμενα προκλήθηκε από μια επιστολή που έστειλε ο βούλγαρος συνάδελφός μου Αντώνη Περβάνουα στην ε, Κομισιόν. Σας διαβεβαιώνω ότι στη Βουλγαρία έχουμε αρμόδιους οργανισμούς δημοσιονομικούς και δημοσιονομικού ελέγχου που τα ελέγξανε όλα. Η δήλωσή μου λοιπόν για τα συμφέροντά μου και θέματα διαμάχης συμφερόντων λοιπά Έχουν, η δήλωσή μου έχει ελεγχθεί από τη Βουλή, από μια επιτροπή ε, σαν τη δική σας εδώ, που αποφάσισε ότι όλα ήταν εντάξει. Και όχι μόνο εντάξει, αλλά τέλεια, τελείως νομότυπα. Αν θέλετε μπορείτε και εσείς να εξετάσετε το φάκελο αυτό, αν θέλετε να σας το στείλω. Εγώ δεν κρύβω τίποτα. Η εταιρεία αυτή, Global Consult δηλαδή, δεν εργαζόταν, δεν λειτουργούσε την εποχή της δήλωσης. Και το δηλώνουν αυτό και οι δημοσιονομικοί οργανισμοί της χώρας μου. Συμπληρωματική, ναι, αν αναμένατε την ερώτηση αυτή, τότε θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα για μας. Θα μας είχατε απαντήσει πιο ουσιοδός. Εγώ ρωτώ, την πουλήσατε την εταιρεία Global Consult και αν ναι, για ποια τιμή. Και αν ναι, επίσης γιατί δεν δηλώθηκε αυτό. Κυρία Γέλεβα. Η εταιρεία είναι δεδηλωμένη ως εταιρεία η οποία όμως δεν εργαζόταν, δεν λειτουργούσε. Δεν ήταν ενεργή στην αγορά. Αυτό φαίνεται από τα χαρτιά μου. Και επειδή το θέμα είναι σημαντικό, θα ήθελα να το απαντήσω στη μητρική μου γλώσσα. Όχι τώρα, όμως σε άλλη ερώτηση. Okay, when then we take extra time. Ε, τότε θα πάρουμε το χρόνο για να το πει στη γλώσσα της, ορίστε. So, I can answer the question. Okay. Uh, бих искала да отговоря uh, на въпрос, uh, понеже вие го задавате. Θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση αυτή. Είναι δεύτερη φορά που μου κάνετε την ίδια ερώτηση. Πρόκειται για ανυπόστατες αιτιάσεις που προέρχονται από τη συνάδελφό μου Αντώνια Παρβάνοβα, Ευρωβουλευτή, η οποία απίφθινε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να σας αποδείξω, να σας δείξω αν θέλετε όλα τα επίσημα έγγραφα που αφορούν αυτό το θέμα. Αν θέλετε μπορώ να σας τα διαβιβάσω. Είμαι σε θέση να το κάνω χωρίς να καταναλώσω περισσότερο χρόνο αυτή τη στιγμή για να μπω σε λεπτομέρειες που πραγματικά ε, σπαταλούν πολύτιμο χρόνο εδώ. Στη χώρα μου υπάρχουν θεσμοί οι οποίοι επιφορτίζονται με τον οικονομικό έλεγχο, λογιστικό έλεγχο και κάθε είδους οικονομικό έλεγχο για να ε, εξασφαλίζουν ότι ε, τηρούνται οι κανόνες της διαφάνειας. και σας απευθύνω έκκληση. Ας συνεχίσουμε εδώ τη συζήτησή μας, την ουσία την ίδια του χαρτοφυλακίου μας μου και σας διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο να σας δείξω, να σας αποδείξω από τα επίσημα έγγραφα τα οποία έχουν δημοσιευθεί από τις αρμόδιες βουλγαρικές αρχές. Όποιος θέλει να έχει περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί να απευθυνθεί σε μένα προσωπικά και να του τις δώσω όποιος θέλει περισσότερες προφορίες να έρθει και στη Βουλγαρία. Να δει την πόλη στην οποία ζω και εργάζομαι, να γνωρίσει το σύζυγό μου αν θέλετε και τις βουλγαρικές αρχές και να ε, βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει τίποτα κρυφό και τίποτα παράνομο. Τώρα νομίζω ότι καλό θα ήταν να επικεντρωθούμε στην ανθρωπιστική βοήθεια. Τόσος κόσμος υποφέρει, χάνει τη ζωή του στον κόσμο. Και εμείς αναλωνόμαστε σε τέτοιες συζητήσεις, με ανυπόστατες αιτίας. Και πάλι επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχει τίποτα παράνομο ούτε στις δικές μου δραστηριότητες ούτε στις δραστηριότητες του συζύγου μου και δεν υπάρχει καμία ε, έρευνα που να έχει ξεκινήσει τη δικαιοσύνη ούτε εναντίον εμού ούτε εναντίον του συζύγου μου ξέρω ποιο σας έδωσε τόσα στοιχεία, τόσες βάσεις, τι σα σωθεί να μου κάνετε τόσες ερωτήσεις και να με εγκαλείτε. Αλλά και πάλι αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι αυτά τα σημαντικά θέματα τη συζήτησή μα σήμερα. Σας ευχαριστώ. Nous reprenons notre tour de questions-réponses et la parole. Συνεχίζουμε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Ο κύριος Σαχραντήλ έχει το λόγο από τους συντηρητικού. Thank you, Madam Chair. Uh, Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν την πρώτη μου, στην πρώτη μου μάλλον παρουσίαση αναφέρθηκα στην επιστημιστική βοήθεια και στην επιστημιστική κρίση και θα ήθελα να ρωτήσω την υποψήφια επίτροπο. Ποια είναι η προτίμησή της, απελευθέρωση του εμπορίου ή νέα πολιτική επιστημιστικής βοήθειας σε περιπτώσεις κρίσεων και έκτακτης ανάγκης. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κυρία Γέλεβα. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση αυτή. Σε διεθνές επίπεδο γνωρίζετε πολύ καλά ότι προσπαθούμε να ε, παρακολουθήσουμε τη μεταρρύθμιση της σύμβασης που αφορά την επιστημιστική βοήθεια και να συνεργαζόμαστε με τρόπο ενεργό και επιμένω σε αυτό εγώ να έχουμε ενεργή συμμετοχή στη συζήτηση αυτή. Τώρα σε επίπεδο επιχειρησιακό συμμετέχουμε πάρα πολύ ε, στη χρήση ε, νέων μεθόδων και νέων ε, τρόπων για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και πιο συνεκτικοί στη δράση μας τόπου. Παραδείγματα θα ήθελα να αναφέρω μερικά μόνο, Φερρυπίν, προσπαθούμε να επιδεικνύουμε καινοτομία και να εφευρίσκουμε νέες δυνατότητες, νέα μέσα, νέα εργαλεία, να μην παρέχουμε μόνο τρόφιμα, αλλά και χρήματα για την αγορά τροφίμων, σε περιπτώσεις ε, που προσπαθούμε επίσης να υποστηρίσουμε τις τοπικές αγορές και τους εγχωρίους ε, εμπόρους. Μπορούμε λοιπόν να επιδεικνύουμε δείξουμε μεγαλύτερη εφευρετικότητα για να διαφοροποιούμε τις μεθόδους παροχής επιστηστικής βοήθειας ε, και να προλαμβάνουμε τέτοιου είδους κρίσεις. Follow-up question. Επόμενη ερώτηση. Έχω ένα διαδικαστικό να θέσω. Μα έχω συμπληρωματική ερώτηση. κυρία Τσίμερ. κυρία Γέλεβα, εδώ είμαι. Μα έχω ένα διαδικαστικό έλεγα. Κοιτάξτε, τώρα έχουμε μια συζήτηση εδώ και γινόμαστε μάρτυρες σε μια συζήτηση όπου χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια, πιστεύω. Ακούστηκε το όνομα μιας βουλευτού, της κυρίας ε, Βάνοβα, ε, η οποία ε, υποτίθεται ότι υποκίνησε τις κατηγορίες τις οποίες συζητούμε και αφορούν την ακαιρεότητα της κυρίας Γέλεβα. Πιστεύω ότι θα ήταν σωστό να δώσετε το λόγο στην κυρία Παρβάνοβα, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να κάνει μια δήλωση σχετικά. Πολύ καλή ιδέα, λέει η Πρόεδρος. Και ως Πρόεδρος της Επιτροπής θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για μια τέτοια δήλωση. Ε, Ευχαριστώ. Μου δίνετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, επειδή ακούστηκε το όνομά μου, παίρνω το λόγο επί του προσωπικού, ότι ενημέρωσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να σας πω ότι ε, εξεδόθη μια ανακοίνωση που μου ζήτησαν ε, να ε, προβώ σε μια ενημέρωση. Αυτά που είπε η κυρία Γέλεβα, φοβούμε, δεν είναι αληθή. Εάν δείτε... Ε, το προφίλ της, το επίσημο που έχει υποβάλει στην Επιτροπή μας, στο Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέρει, είναι ε, στο βιογραφικό της το επίσημο ότι έχει δραστηριότητες στην εταιρεία αυτή από το 2001 έως το 2003 και στη συνέχεια από το 2004 ως συγγνώμη, 2006 διορθώνει μιλήτρια ως 2007. Αυτό δεν συνάδει όμως με τους κανόνες για τις, από 14 Ιουνίου 2006 μέχρι τις 9 Απριλίου 2009 ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Υπάρχει όμως βουλγαρική νομοθεσία που ορίζει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ε, υπάρχει ασύμβατο και ασυμβίβαστο με τη βουλευτική ιδιότητα ή την ιδιότητα του Ευρωβουλευτού. Δεν μπορεί να κατέχει τέτοια θέση σε τέτοιες εταιρείες. Επιπλέον, επολύθη η εταιρεία αυτή μεν, αλλά όχι ακριβώς, έχει αλλάξει όνομα και παραμένει η ιδιοκτησία στο 60% στα χέρια της κυρίας Γέλεβα. Αυτά είναι επίσημα στοιχεία τα οποία ελάβαμε και τα οποία ε, ανέλησε και δικηγόρος. Επίσης, σήμερα είδα να δημοσιεύεται αυτό στους Financial Times και ε, είναι δημόσια, δεν είμαι εγώ εκείνη που ε, τα δημοσίευσα, δεν έκανα τίποτα κακό. Απλώς έδωσα αυτές τις πληροφορίε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αποφύγουμε ε, οποιαδήποτε μελλοντικά λάθη. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Παρβάνοβα. Η κυρία Γέλεβα. You have the floor to answer this observation, this very Έχετε το λόγο για να απαντήσετε σε αυτές τις πολύ σημαντικέ παρατηρήσει. Διότι αν σας ε, εννοήσα σωστά, δεν μιλούμε για φήμε, αλλά για επίσημα έγγραφα και στοιχεία που δείχνουν ότι η δήλωση της υποψηφίας επιτρόπου δεν συνάδει με τη βουλγαρική νομοθεσία. Αυτό δεν μας λέτε. Οπότε, κυρία Γέλεβα, παρακαλώ. σα σας όσο χρόνο έδωσα και στην κυρία Παρβάνοβα για να απαντήσετε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ούτε εγώ, ούτε η κυρία Περβάνοβα είμαστε νομομαθείς. Γι' αυτό λοιπόν επαναλαμβάνω και τονίζω. Έχω ένα φάκελο με όλα τα στοιχεία, με όλα τα απαραίτητα έντυπα και αυτός ο φάκελος δείχνει ότι σέβομαι τη βουλγαρική νομοθεσία. Ελπίζω ότι η Επιτροπή σας θα συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος που μας έφερε εδώ. Οι συνεργάτες μου θα σας μοιράσουν το φάκελο αυτό. Θέλω να σας πω μόνο ότι αυτή η επιχείρηση που αναφέρθηκε κατ' επανάληψη, αυτή η εταιρεία είναι ανενεργή. Εδώ και πολλά χρόνια είναι ανενεργή. Και με βάση τη βουλγαρική νομοθεσία ε, αυτό το πράγμα έχει δηλωθεί και μπορώ να το αποδείξω και βάση τεκμηρίων. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να επαναλαμβάνω αυτά τα πράγματα ιστοδυνικές. Δεν ξέρω ποιες είναι οι συνήθεις πρακτικές στην Επιτροπή σας. Δεν ξέρω αν ε, συνηθίζετε να ακούτε τέτοιες δηλώσεις, αλλά θα ήθελα να σταματήσουμε και να λάβετε υπόψη σας τα έγγραφα. Υπάρχουν τα έγγραφα. Εάν είχα παραβιάσει την ε, νομοθεσία, οι βουλγαρικές αρχές θα το είχαν διαπιστώσει και θα το είχαν δημοσιοποιήσει. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας διαβεβαιώσω ότι τα δικαστήρια στη χώρα μου και οι οικονομικές αρχές λειτουργούν. Υπάρχουν όλοι οι απαραίτητοι θεσμοί για να αποφασίσουν και να πιστοποιήσουν την, το γνήσιο των εγγράφων αυτών. Υπάρχει μάλιστα και μία επιτροπή ανάλογη με τη δική σας που ασχολήθηκε με το θέμα. Σήμερα νομίζω ότι έχουμε συγκεντρωθεί εδώ για να σας παρουσιάσω τις απόψεις μου σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια. Επαναλαμβάνω ότι η Βουλγαρική Κοινοβουλευτική Επιτροπή δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία σύγκρουση συμφερόντων. Θα σταματήσουμε εδώ γιατί σας δώσαμε τον ίδιο χρόνο που δώσαμε στη μάρτυρα, λέει η Πρόεδρος, ε, και ε, θα ζητήσουμε να διαβιβαστεί ο φάκελος ε, δήλωση οικονομικών συμφερόντων της κυρίας Γέλεβα για να τον εξετάσουμε επίσης. Κυρία Πρόεδρε, δικαστικό. Παρακαλώ, κύριος Μίτσελ. Ο οικονομικός ελεγκτής ε, έχει ως στόχο πραγματικά να επαγρυπνεί και όχι να επιτίθεται. Έκανε μια δήλωση η κυρία Γέλεβα, ε, θα πρέπει να ελέγξουμε ε, ε, το κατά πόσο η κυρία Γέλεβα είναι ικανή και σε θέση να λάβει αυτό το χαρτοφυλάκιο, αν αυτά που δηλώνει για το οικονομικό της ε, ε, συμφέρον θα τα θεωρήσουμε ότι δεν μας ικανοποιούν, να το δούμε αργότερα. Αλλά μια τέτοια διαδικασία είναι λάθος. δεν είναι σωστό ε, ε μέσω μια ερεύνης να κυκλοφορούν και διανέμονται διάφορα μονομερί, μονόπλευρα έγγραφα. Δεν χρειάζεται τώρα να εξετάζουμε διάφορα έγγραφα προς αυτή την κατεύθυνση κατά τη διάρκεια της συνεδρίας τη Επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Ναι. ναι c'est, elle n'est pas là. Mad... Non. Oui, c'est ça. Nous passons maintenant à l'audition de la commission associée. Τώρα περνάμε στην ακρόαση των υπολείπων επιτροπών που συμμετέχουν στη διαδικασία. Έχετε και εσείς διαδικαστικό. Ναι, διαδικαστικό κύριε Πρόεδρε. Λέει ο κύριο Λάγκεν. Διανέμονται διάφορα έγγραφα αυτή τη στιγμή στα γερμανικά και στα βουλγαρικά, αμετάφραστα. Και μόνο μερικά μέλη τα λαμβάνουν. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα κατά τη διάρκεια της ακρόασης. Δεν μπορούμε να μοιράζουμε έγγραφα μη μεταφρασμένα και ε, να κάνουμε διακρίσεις. Παρακαλώ αυτό να το διακόψετε και να συλλέξετε και πάλι όλα τα έγγραφα που έχουν μοιραστεί. Je vais donner raison à cette demande. Δίκιο. Θα ήθελα τα κείμενα τα οποία έχουν διανεμηθεί να τα μαζέψουν οι κλητήρες παρακαλώ. Τώρα κυρία Τσίμερ. Ας περάσουμε στις ερωταποκρίσεις. Έχετε 45 δευτερόλεπτα, κυρία Τσίμερ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ είχα πάρα πολλές ερωτήσεις ε, επί της ουσίας για την κυρία Γέλεβα σε σχέση με το αντικείμενό της και πώς θα ασκήσει τα καθήκοντά της. Αλλά τώρα διαπιστώνω και εγώ δυστυχώς ότι δεν μπορώ να διαχωρίσω τα δύο πράγματα. Ε, το αίτημα για διαφάνεια στην Επιτροπή μας, η δυνατότητα λήψη αποφάσεων από εμά, δηλαδή τα μέλη της ε, Επιτροπής μας για να κάνουμε μια πρόταση, μια αιτιολόγηση προς τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, ε, διακυβεύονται και η ικανότητα διάκρισης μας. Γι' αυτό από ασύρω ε, την ερώτηση που θα είχα και ζητώ να διευκρινιστούν τα πράγματα σε σχέση με την κυρία Γέλεβα και προς το δικό της συμφέρον και να αναβληθεί η ακρόαση μέχρι να επανέλθει ένα κλίμα ηρεμίας για να μπορέσουμε σωστά να προχωρήσουμε στην ακρόαση αυτή. Euh, Εντάξει, μου φαίνεται ότι συνεχώς το ίδιο θέμα πανερχόμαστε και ίσως αυτό πρέπει να το λύσουν οι συντονιστέ και συντονίστριε. Είναι τεχνικό θέμα. Θέλετε κυρία Τσίμερ να το θέσετε τεχνικά. Ε, τότε... Ναι, αλλά θέλω να έχουμε ένα κλίμα ήρεμο για να μπορούμε να έχουμε σωστές ερωτήσεις και απαντήσεις με νόημα. Στο, επί της ουσίας θέλω να μάθω από μια μέλουσα επίτροπο τι θέλει να κάνει για να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι με την κλιματική αλλαγή έχουμε όλο και πιο συχνές θεομηνίες και πώς μπορούμε να προλάβουμε αυτές. Και ρωτώ, τι γίνεται με την πρόληψη ή με την ε, ε, μετρίαση των ε, συνεπειών το βλέπει ως αντικείμενο του δικού της χαρτοφυλακίου και ε, θέλει να δημιουργηθεί μια ξεχωριστή διευκόλυνση οικονομική για την αντιμετώπιση αυτών των κρίσεων. Κυρία Γέλεβα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Τσίμερ για την ερώτησή σας, απάντως στα γερμανικά. Και θυμόμαι και την καλή συνεργασία που είχαμε στην Κοινωνική Επιτροπή κατά τη διάρκεια της θητείας μου εδώ ως Ευρωβουλευτού και θα ήθελα να σας πω το εξής το ερώτημα που θέτεται αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προηγουμένως, στις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις είπατε τι γίνεται με την τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με ρωτήσατε. Έτσι, αν μπορούμε να συνεργαστούμε και αν έχουμε πραγματικά εργαλεία διαφορετικά για την πολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Όπως γνωρίζετε, αυτό τον καιρό είναι πάρα πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε αλλάζοντας τα μέσα και τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Και εδώ πιστεύω ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων μας θα είναι και αυτό. Και πραγματικά προσβλέπω στις προτάσεις του Κοινοβουλίου για μια καλή συνεργασία, έτσι ώστε να αναπτύξουμε νέες δυνατότητες και να αξιοποιήσουμε νέες ε, δυνατότητες και από τα κράτη-μέλη, αλλά γιατί όχι και από θεσμικά ιδρύματα που αναφέρατε κι εσείς, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, να βρούμε χρήματα ε, για να κάνουμε κάτι στον προπολογισμό μας για την ανθρωπιστική βοήθεια. Προς το παρόν όμως αυτό είναι μόνο περιορισμένο, το γνωρίζετε και εσείς ως δυνατότητα, μπορούμε να το αξιοποιήσουμε στο μέλλον. Και να αλλάξουμε μεταξύ άλλων και την νομική βάση, την νομοθετική βάση για να είναι πιο εύκολα και πιο ταχαία όλα αυτά. Έχει καταφτάσει η κυρία Νικόλ Σινκλέρ, όχι. Τότε θα ήθελα να δώσω το λόγο στην ε, στην δεδεμένη Επιτροπή Περιβάλλοντος που έχει προσκληθεί. Ο κύριος Σκυλακάκης, παρακαλώ. Madam Zaleva, here. Here, here, here. Ε, natural disasters have been escalated. Οι θεομηνίες αυξάνονται τα τελευταία χρόνια και χειροτερεύουν λόγω των κλιματολογικών αλλαγών, όπως το είπατε κι εσείς. Υπάρχουν θέματα όπως οι πυρκαγιές των δασών στην νότια ιδίω Ευρώπη, όπου τα πράγματα χρόνο με το χρόνο χειροτερεύουν. Και αυτό μάλλον συνδέεται με τις κλιματολογικές αλλαγές. Τι σκοπεύετε να κάνετε ώστε οι κοινοτικοί μηχανισμοί για την πολιτική προστασία να είναι πιο αποτελεσματικοί, ιδιαίτερα όταν είναι πολλαπλές οι θεομηνίες αυτού του είδους. Κυρία Γέλεβα, Ευχαριστώ για το ερώτημα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να θυμηθούμε πόσες πολλές πυρκαγιές σημειώθηκαν φέτος και στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις θα συνεχίσουν τέτοιες πυρκαγιές και θα αντιμετωπίσουμε παρόμοιες θεομηνίες και γι' αυτό θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης μπορούμε να κάνουμε μερικά πράγματα για να αντιμετωπίσουμε, να βελτιώσουμε τις δυνατότητές μας ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να επιδείξουμε περισσότερη αλληλεγγύη. Πρώτον, έχουμε στη διάθεσή μας το πειραματικό ή πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο θα αναθεωρηθεί, θα αξιολογηθεί σε λίγο για τη χρησιμοποίηση Καναντέρ σε περιπτώσεις πυρκαγιάς των δασών. Αλλά πέρα από το πειραματικό ή πιλωτικό πρόγραμμα πρέπει να δώσουμε περισσότερες δυνατότητες στα κράτη-μέλη να χαρτογραφήσουν, να δουν, να αναλύσουν τα πράγματα για να έχουμε μια σαφή γνώση τι μέσα διαθέτουμε στην περίπτωση δασικής πυρκαγιάς. Πρέπει να ενδυναμωθεί η συνεργασία και μεταξύ των χωρών μελών αλλά και μεταξύ χωρών και κομισιών. Και αν όντως οριστώ στη θέση αυτή, από το Κοινοβούλιο, αν εγκριθεί ο διορισμός μου, είμαι διατεθειμένη να ενδυναμώσω τις δυνατότητες και την προετοιμασία. Τελείωσε ο χρόνος στη συμπληρωματική. Δύο λόγια μόνο. Ο προηγούμενος ε, αρμόδιος επίτροπος είχε πει ότι το πιλωτικό επιρωματικό πρόγραμμα είναι απαραίτητο γιατί χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει τίποτα. Θέλετε λοιπόν να το αναθεωρήσετε ή να το επεκτείνετε κιόλας. Κύριε κυρία Βά. Πρέπει να δούμε πρώτα τι θα πει η ανάλυση και μετά θα, με τη βοήθεια και της Επιτροπής σας και άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών όπως η Επιτροπή Περιβάλλοντος θα μπορέσουμε να δούμε τα πράγματα καθαρότερα και σαφέστερα αν χρειάζεται δηλαδή αναθεώρηση ή επέκταση. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και πολλές δηλώσεις του Κοινοβουλίου είναι σαφέστατες αρχίζει εδώ ο δεύτερος γύρος ερωτήσεων. Ο λόγος στον κύριο Κασμάρεκ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Επίτροπε, βασιστήκατε ιδιαίτερα σε θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας και προγράμματα αντιμετώπισης κρίσεων και θεομηνιών. Τι άλλο αποτελεί τμήμα της εντολής σας για την ανθρωπιστική βοήθεια εκτός από αυτά που αναφέρατε ήδη. Ορίστε κυρία Γέλεβα. Ε, βέβαια, καταρχήν η αναθεώρηση του προγράμματος δράσης που προχωράει πολύ καλά. Έχουμε 42 μέτρα αναλύσει ή εφαρμόσει μάλλον ήδη Και θα έλεγα ότι σαφές μήνυμα που, ήθελα, που θέλω να σας δώσω είναι ότι το έγγραφο αυτό, η μελέτη αυτή είναι πολύ καλά προετοιμασμένη, συνυπογράφεται και από τα τρία θεσμικά όργανα, αλλά υπάρχει χώρος για βελτίωση φυσικά. Το σεβασμό δηλαδή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και τις σχέσεις πολιτικών και στρατιωτικών δυνάμεων καθώς και τις επιπτώσεις, τις ανθρωπιστικές επιπτώσεις των κλιματολογικών αλλαγών και άλλα. Με τη βοήθεια της Επιτροπής σας και του Κοινοβουλίου ολοκλήρου νομίζω ότι θα μπορέσουμε να προοδεύσουμε σε πολλά από αυτά τα θέματα. Συμπληρωματική. Όχι. Τότε ο κύριος Μπέρμαν. Ευχαριστώ πρόεδρε δεν ικανοποιηθήκα πολύ από τις απαντήσεις σας για τη διαφάνεια που είναι απαραίτητη ποιότητα για έναν επίτροπο. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι το τεχνικό. Τι φρονείτε για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ανθρωπιστικές καταστρο... στην ανθρωπιστική καταστροφή στον κόλφο του Άντεν. Στον κόλπο. κόλπο. Αγέλεβα. Δεν κατάλαβα καλά την τελευταία πρόταση. Μπορείτε τι φρονείτε για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίλυση της ανθρωπιστικής κρίσεως στον κόλπο του Άντεν. Άντεν. Πρέπει να είμαστε πολύ δραστήριοι επιτόπου και η ανθρωπιστική βοήθεια όπως ξέρετε είναι κάτι το απαραίτητο και πρέπει να χορηγείται επί τόπου. Έχουμε εμπειρογνώμονες, επαγγελματίες και αν με διορίσει το κοινοβούλιο θα ήθελα να πάω να δω η ίδια με τα μάτια μου πώς έχει η κατάσταση εκεί και σας διαβεβαιώνω ότι για πολλές τέτοιες καταστάσεις και κρίσεις όπως αυτή που αναφέρατε θα πάω να επισκεφθώ τα πράγματα αυτοπροσώπως και να δω τι γίνεται. Συμπληρωματική. Σε μια χώρα σαν τη Σομαλία είναι πολύ δύσκολο να παραμείνει κανείς αδέκαστος και ουδέτερος. Τι θα κάνετε, πώς θα δράσετε. Σε πολλές χώρες είναι δύσκολο να διατηρήσει κανείς τον αδέκαστο και ουδέτερο χαρακτήρα που πρέπει να έχει χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά αυτές είναι οι αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας και όσο δύσκολο και να είναι, αν υπάρχει συνένεση, όλα γίνονται. Αυτό θα ζητήσω λοιπόν και σε χώρες σαν τη Σομαλία και σε άλλες. Θα προσπαθήσω και θα ξαναπροσπαθήσω με κάθε τρόπο να πείσω τις τοπικές αρχές να μας δώσουν τη δυνατότητα, την πρόσβαση για να χορηγήσουμε ανεξαρτήτως ανθρωπιστική βοήθεια. Ο κύριος Γκέρεντς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι προφανές ότι η Ένωση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη χορήγηση για διεθνού ανθρωπιστική βοηθεία και αυτό αναγνωρίζεται και από τον ΟΗΕ. Θέλετε λοιπόν να δώσετε κάποια νέα πολιτική ορμή για την α, μεταρρύθμιση της λειτουργίας του ΟΗΕ για να προσαρμοστεί αυτή η λειτουργία καλύτερα στις σημερινές συνθήκες, κυρία Γέλεβα έχει το λόγο. Στο ο ΟΗΕ και όλοι οι άλλοι διεθνείς οργανισμοί είναι σημαντικό τμήμα του δικτύου μας ανθρωπιστικής βοηθείας. Μεταξύ άλλων και οι μη κυβερνητικές και ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός και άλλες. Πρέπει όμως να γίνει και η μεταρρύθμιση της λειτουργίας του ΟΗΕ, συμφωνώ, συμφωνώ, αλλά δεν έχω έτοιμη πρόταση γιατί μόνο διάλογο μπορούμε να κάνουμε με τον ΟΗΕ, όχι να τους δώσουμε εντολές και καλύτερο συντονισμό να ζητήσουμε συνδυασμό με τις δικές μας προσπάθειες δηλαδή να τους βοηθήσουμε, όχι να τους καθοδηγήσουμε, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και τη δυνατότητα με την εντολή μου, διεθνής συνεργασία δηλαδή μεταξύ άλλων, να είμαστε πιο δραστήριοι σε συνεργασία με την Κατερίνα Άστον και άλλους επιτρόπους έτσι ώστε να υπάρξει μια πιο αποτελεσματική και διαφανής λειτουργία και για τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ. συμπληρωματικό κύριε Γκέρντς. Όχι. Από τώρα και στο εξή δεν θα γίνονται συμπληρωματικέ γιατί έχουμε καθυστερήσει υπερβολικά. Δυόμιση λεπτά και όχι τρισήμιση λοιπόν οι ερωταπαντήσει. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Σερσέντ. Να πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Γελέβα, εγώ έχω προετοιμαστεί. Δεν θα θέσω ερωτήματα για την βουλγαρική νομοθεσία, αλλά για τις αρχές που έχουμε εδώ στην Ένωση. Ένα πολύ απλό ερώτημα. Έχω εδώ πέρα χαρτιά για την Global Consult και μια άλλη εταιρεία με το όνομά σας. Την Global Consult την πουλήσατε, αλλάξατε το όνομά της, είστε ακόμη ιδιοκτήτριά της ή του Ότος Πάρ. Ευχαριστώ. Είπαμε ότι το θέμα αυτό θα το λύσουν οι συντονιστές και οι συντονίστριες. Μα κυρία Πρόεδρε μου, η κυρία Κέλεβα δεν είναι προετοιμασμένη να απαντήσει σε τέτοια ερωτήματα, αλλά θα έπρεπε, είπε ότι τα ανέμενε. Εγώ γιατί ετοιμάστηκα. Έχω προετοιμαστεί και για ερωτήσεις ανθρωπιστικής βοηθείας αλλά ούτε αυτές απαντήθηκαν. Και αν δεν είναι προετοιμασμένη η υποψήφια επίτροπος δεν μπορώ και εγώ να θέσω το ερώτημά μου. Αυτό είναι περίπου πολύ περίεργος τρόπος να ζητάμε διαφάνεια εδώ μέσα. Παρακαλώ κυρία Γελέβα, απαντήστε μου αυτή την απλή ερώτηση που έκανα. Για η τελευταία φορά. Κυρία Γέλεβα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν είμαι ιδιοκτήτρια της Global Consult. Ούτε και της άλλης εταιρεία με το άλλο όνομα. Δεν είμαι ιδιοκτήτρια. Δεν ξέρω που βρήκατε αυτά τα στοιχεία. Σας παρακαλώ, ας επικεντρωθούμε στο θέμα μας. Και, εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε και τα βουλγαρικά μητρώα. Σας προσκαλώ, ελάτε σε μένα. Ελάτε μαζί μου στη Βουλγαρία και να τα δείτε όλα οι όμασης. μπορείτε να δείτε οποιοδήποτε και να τσεκάρετε οποιοδήποτε αρχείο θέλετε. Είμαι από τον Μπούργκας. Από εκεί προέρχεται αυτό. Υπάρχει συγκεκριμένο αρχείο, από εκεί προέρχονται αυτά τα στοιχεία που έχω συγκεντρώσει. Νομίζω ότι λειτουργούν ε, οι αρχές πολύ καλά. Υπάρχει αυτό το αρχείο, είναι στη διάθεση τη δική σας και όλων εδώ, όλων των υπόλοιπων ευρωβουλευτών. Επαναλαμβάνω η τελευταία φορά, δεν είμαι ιδιοκτήτρια. Δεν είμαι. Ούτε της Global Consult, ούτε της άλλης εταιρείας που δεν συγκράτησαν καν, που δεν καν το όνομα. Είσαστε έτοιμοι να ταξιδέψετε μαζί μου στη Βουλγαρία σας έχω προσκαλέσει. Θα συνεχίσουμε τώρα, είπε η Πρόεδρος. Ο κύριος Σαχαντρίλα. 45 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ας ξαναπάμε στην ανθρωπιστική βοήθεια. Υπάρχει μια μονάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θαυμάσια μονάδα, ε, European Commission Emergency Aid το ΕΚΟ. Υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια που έχετε σκεφτεί, ούτως ώστε αυτή η μονάδα να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά. Ακόμα. Παραδείγματο χάρη, έχετε κάποια σχέδια για να δημιουργηθούν στρατηγικά αποθέματα ανά τον κόσμο. Κυρία Γέλεβα, έχετε τον λόγο. Είμαι έτοιμη να συνεργαστώ με όλες τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συνεργασία είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Η δουλειά που κάνουμε είναι επιχειρησιακή σε μεγάλο βαθμό. Δίνουμε βοήθεια και μειώνουμε τα δεινά που αντιμετωπίζουν οι πληθυσμοί σε διάφορες χώρες του πλανήτη. Ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Προτιμώ να έχουμε καλύτερο συντονισμό και καλύτερο διάλογο μεταξύ των υπηρεσιών. Η μακροπρόθεσμη προετοιμασία επίσης είναι πολύ σημαντική για να είμαστε πιο προετοιμασμένοι, ακόμη πιο προετοιμασμένοι για τις κρίσεις. Ανέφερα ήδη ότι θα ήθελα να ετοιμάσω και διάφορα σενάρια πριν να ξεσπάσουν οι κρίσεις, οι ενδεχόμενες κρίσεις. Κυρία Στρίφλερ, κυρία Γέλεβο, για να μην μπερδέψουμε το ρόλο και την ταυτότητα μεταξύ των ανθρωπιστικών οργανώσεων και των στρατιωτικών οργανώσεων, ε, η συνένεση για τις ανθρωπιστικές οργανώσεις θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το ρόλο που έχει ο καθένας από τους εταίρους και να μην ξεχνάμε ε, το Όσλο και τις κατάλληλες οδηγίες. Θα πρέπει να υπάρχει ανεξαρτησία, αμεροληψία. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να υπάρχει συνένεση σε αυτό το σημαντικό τομέα, ειδικά στο Αφγανιστάν. Πώς θα ενδυναμώσετε το διάλογο με τους στρατιωτικούς φορείς και τους πολιτικούς ε, στα πλαίσια της μιας οποιασδήποτε ανθρωπιστικής επιχείρησης. Κυρία Γέλεβα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση. Και είναι προτεραιότητά μου η σχέση μεταξύ των ανθρωπιστικών οργανώσεων και των στατιωτικών δυνάμεων. Πρέπει να μην υπάρχει σε καμία περίπτωση σύγχυση ανάμεσα στο ρόλο και την εντολή των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και στρατιωτικέ δυνάμει και οργανώσεις. Για το Αφγανιστάν που αναφέρατε. Είναι κακό παράδειγμα, όντω. Όπου η αρχή της ανεξαρτησίας δεν έχει γίνει σεβαστή. Έχουμε όμως και ένα καλό αντιπαράδειγμα στο Τσάντ. Αυτό που σκοπεύω να κάνω είναι να ενδυναμώσω φυσικά το διάλογο σε ένα πρώτο επίπεδο μεταξύ των στρατιωτικών δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και ε, διάλογο με τους Υπουργούς Εξωτερικών και Υπουργούς Άμυνας, προκειμένου να ξεκαθαρίσουν οι... τα όρια ανάμεσα στο ρόλο και την εντολή των στρατιωτικών δυνάμεων και των ανθρωπιστικών δυνάμεων και οργανώσεων. Επίσης θα ήθελα να έχω έτοιμα σενάρια πριν ληφθούν οι πολιτικές αποφάσεις για στρατιωτική δράση. Και τώρα ένα μέλος της Εξωτερικής Επιτροπής ε, εκπροσωπείται η Επιτροπή αυτή τον κύριο Πάσκου η Επιτροπή Άθλητη Εξωτερικών Υποθέσεων. Σας ευχαριστώ. Με τις συζητήσεις αυτές που γίνονται τώρα, α, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις ε, στη δουλειά σας. Μία πρόληψη, η μία αντίδραση και η τρίτη συνδυασμός των δύο. Πώ σκοπεύετε να συνδυάσετε τις δύο πρώτες, κυρία Γέλεβα. Uh, Θα έχουμε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση και τα τρία στοιχεία. Είναι κάτι που προκύπτει ξανά και ξανά στη συζήτησή, μας, συζήτησή μας, ότι πρέπει να είμαστε δραστήριοι, ενεργητικοί. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, Φερρυπίν, Το τρίτο πυλώνα, ε, την πρόληψη των ε, φυσικών καταστροφών. Τρίτος πυλώνας για την ανθρωπιστική βοήθεια. Και περιέχει πολλά στοιχεία που μας επιτρέπουν να λειτουργήσουμε και να προωθήσουμε την πρόληψη. Το θέμα είναι όχι μόνο να έχουμε γρήγορη απόκριση, αλλά πρόληψη, δηλαδή κατάρτιση, άσκηση, εμπλοκή νέων εταίρων στο πλευρό μας μέσα σε συνθήκες διαφάνειας. Όλοι να γνωρίζουν τα μέσα που έχει στη διάθεση του άλλος. Να προσπαθήσουμε να κοινοτοποιήσουμε και να αναλύσουμε εκ των προτέρων διάφορα σενάρια για κρίσεις. Έχουμε την ευθύνη, έχουμε και το δυναμικό για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι υπάρχει η προσθέμενη αξία από το συνδυασμό αυτών των προσπαθειών. Το συνδυασμό στα πλαίσια ενός χαρτοφυλακίου. Ε, συμπληρωματική ερώτηση, όχι, δεν υπάρχει. Και τώρα έχουμε την ε, σύνοδο του follow-up, έξι λεπτά θα Αλλά δεν έχω λάβει ερωτήσεις από τις πολιτικές ομάδες, άρα δεν θα λάβει χώρα. Επομένως, εντάξει, είμαστε μέσα στο χρονοδιάγραμμά μας. Και μπορούμε να επανέλθουμε ε, στι ρωτοποκρίσεις των 3,5 ε, λεπτών. Κυρία Κρετού, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Στην ε, Επιτροπή περιβάλλοντος ε, θα θέλαμε να θέσουμε ερώτηση για τις ε, πυρκαγιές στην Νότια Ευρώπη. Υπάρχουν και τα προβλήματα των πυρκαγιών ε, που ξεπερνάνε τα σύνορα. Μας δώσατε μέρη στην εισαγωγή σας μία απάντηση, όπου είπατε ότι υποστηρίζετε ένα νέο ευρωπαϊκό σώμα για την πολιτική προστασία. Πώς θα πείσετε την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να δώσουν κονδύλια για αυτό το νέο φορέα πολιτικής προστασίας στην Ευρώπη. Λαμβάνοντα υπόψη ότι ήδη είναι δύσκολο να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας που έχουμε δώσει προς τις πιο φτωχέ χώρες. Έχετε το λόγο, κυρία Γέλεβα. Ε, ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση, πολύ ενδιαφέρουσα. Από το 2006 έχει ξεκινήσει η συζήτηση και καλά κρατεί Ξεκινήσαμε και χάρη στο Κοινοβούλιο ε, ένα καλό πρόγραμμα και χάρη στις επικοδομητικές συζητήσεις που έχουμε μαζί σας για αυτό το θέμα. Μπορούμε να ενδυναμώσουμε τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Και να τα βοηθήσουμε να είναι πιο έτοιμα. Με τη χαρτογράφηση και με την ανάλυση, με την ε, καταλογοποίηση των ε, στοιχείων που έχουν στη διάθεσή τους, ε, του εξοπλισμού και του μηχανισμού που έχουν για να αντιμετωπίσουν τα κατεπήγοντα. Για τις ε, δασικές πυρκαγιές προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε το περασμένο καλοκαίρι αυτά τα αεροπλάνα. Ήταν μια χρήσιμη εμπειρία. Καταρχάς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι πόρους έχουμε στη διάθεσή μας. Και συνεχεία μπορούμε να ζητήσουμε περισσότερους πόρους, μπορούμε να κάνουμε έκκληση για περισσότερους πόρους, γιατί ζούμε σε ισχνές αγελάδες και δεν μπορούμε έτσι εύκολα, έτσι αστόχαστα να ζητάμε περισσότερα. Κυρία Κρέτου, έχετε δεύτερη ερώτηση συμπληρωματική. Σας μίλησα για το νέο σώμα που δεν υπάρχει ακόμα. Θα είσαστε ο υπεύθυνο επίτροπος ε, αυτού του νέου σώματος για την πολιτική προστασία. Γι' αυτό σας ρώτησα. Αυτό το σώμα, έχετε δίκιο, δεν υπάρχει ακόμα. Έχουμε μόνο ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Προσπαθούμε να δούμε αν έχει νόημα να στηθεί αυτό το σώμα. Όταν ολοκληρωθεί το, η πιλωτική φάση, το, συμβούλιο, το Κοινοβούλιο συγγνώμη, θα δώσει τη γνώμη του για αυτό το ζήτημα. Πάντως μην ξεχνάμε ότι η πολιτική προστασία είναι καταρχήν εθνική αρμοδιότητα. Ο κύριος Λουί Μισελ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, υποψηφία Επίτροπε, ε, σύντομα, ποια εργαλεία θα μπορούσατε να προτείνετε για να προωθήσετε την ενίσχυση και κυρίως το σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που καταπατείται και παραβιάζεται χωρίς να έχει την πολιτική δυνατότητα να αντιδράσει η Ευρώπη ούτε καν να καταγγείλει τα φαινόμενα αυτά. Βλέπετε κάποια δυνατότητα σύνδεσης του θέματος αυτού σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ως παράδειγμα. Δεύτερον, κατανοώ ότι θέλησή σα να συνεργαστείτε στενά με τι υπηρεσίε του ΟΗΕ και βεβαίω συμφωνώ. Θα ήθελα όμως να σας ερωτήσω πώς θα το κάνετε αυτό χωρίς να περιορίσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα ρόλο θηρίδας διανομής, ε, μπανάλ, χωρίς ε, ειδική προβολή και ειδική παρουσία. Uh, ευχαριστώ κύριε Μισελ. Καταρχάς σας ευχαριστώ που θέτετε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Ε, κοιτάξτε, εσείς γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε άλλα μέσα, ούτε άλλα εργαλεία από την υγιή διπλωματία για να πείθουμε ε, τις ε, ντόπιε αρχές, τι πολιτικές αρχές να δίνουν ε, πρόσβαση στι ανθρωπιστικέ μας αποστολέ. Μία όμως που αναφέρεται εργαλεία, ε, θα ήθελα να πω εγώ ε, ότι όχι κατά παράδοση, αλλά κάτι που χρησιμοποιείται στην πράξη είναι το μέσο σταθερότητας και κάποια άλλα μέσα που έχουμε στη διάθεση μας στην διεύθυνση ρέλεξ εξωτερικών σχέσεων. Επίσης και στα διεθνή φόρα μπορούμε να ζητήσουμε να γίνεται καλύτερα σεβαστώ το ε, διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε δε ότι ο σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου είναι πάρα πολύ σημαντικός και για ε, την ασφάλεια, την ακαιρεότητα των εργαζομένων στις ανθρωπιστικές οργανώσεις ε, για τη δράση τους και την πρόσβαση στις περιοχές αυτές. Και τέλος, και για την αποτελεσματικότητα των δράσεών μας των ίδιων. Είμαι υπέρ λοιπόν αυτής της προσέγγιση. Έχετε συμπληρωματική ερώτηση κύριε Μισελ. Η κυρία Λεβάιν. Ευχαριστώ. Κυρία Γέλεβα. Λέει κυρία Λεβάιν. Πώς προτίθεστε να εφαρμόσετε αποτελεσματικά τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των θεομηνιών χωρίς ε, περισσότερα χρήματα. Η κλιματική αλλαγή λέμε ότι είναι ανθρωπογενή. Εσείς τι μέτρα θα πάρετε για να προσπαθήσετε να επηρεάσετε τη διεθνή συνεργασία τη αναπτυσσόμενης χώρες για να προληφθούν οι θεομηνίε στη ρίζα του. για παράδειγμα, σκέφτομαι εδώ ότι η λαθρέα υλοτόμηση. Ε, κυρία Γέλεβα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Η κλιματική αλλαγή όντω είναι ανθρωπογενή και όχι θεομηνία. Ανθρωπομηνία. Αλλά δεν είναι ξεχωριστή αρμοδιότητα της ανθρωπιστικής ε, δράσης. Δεν μπορούμε και να παίρνουμε αποφάσεις στο τομέα αυτό, γιατί όπως είπατε δεν έχουμε επιπλέον οικονομικούς πόρους. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αυξήσουμε τη συνειδητοποίηση και να προσπαθήσουμε πραγματικά να είμαστε ενεργοί και δραστήριοι στο πολιτικό επίπεδο, στον πολιτικό διάλογο. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ως υπουργό Εξωτερικών της Βουλγαρίας ήμουν παρούσα στην Κοπενχάγη και παρακολούθησα και τις συζητήσεις και τις εργασίες της. Βεβαίως μπορούμε να είμαστε πιο ενεργοί στις τρίτες χώρες, αλλά γνωρίζουμε ότι έχουν και οικονομικά προβλήματα και δεν ε, είναι σε θέση να συμμετέχουν οικονομικά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι η ανθρωπιστική βοήθεια είναι ένας μόνο τρόπος να βοηθάμε τους ανθρώπους. Δεν είναι η λύση πανάκια για κάθε δεινά, για πάσα νόσο και παν πρόβλημα. Κυρία Λόβιν, έχετε σημαντική ερώτηση. Όχι. Ναι. Είπατε ότι διατελέσετε υπουργό εξωτερικών της Βουλγαρίας. Μπορείτε λοιπόν να μας κάνετε κανένα σχόλιο για το γεγονό ότι δεν παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια η Βουλγαρία. Ναι, ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Όταν ανέλαβα και για μένα σε κάποιο βαθμό αποτέλεσε έκπληξη το γεγονός ότι δεν υπήρχε ανθρωπιστική βοήθεια. Ότι δεν υπήρχε ξεχωριστή υπηρεσία στο Υπουργείο για αυτό το σκοπό. Αλλά πρέπει να σας πω ειλικρινά ότι είναι νέο ζήτημα αυτό ναι. για όλα τα νέα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ε, στο εξάμεινο που ε, ήμουν στο Υπουργείο κατάφερα να δημιουργήσω ξεχωριστή μονάδα στο Υπουργείο Εξωτερικών και για την αναπτυξιακή πολιτική και για την αναπτυξιακή βοήθεια. And, uh, uh, it is uh, really Και είναι πραγματικά πολύ σπουδαίο για μας να γνωρίζουμε ότι όλα τα νέα κράτη-μέλη στην Ένωση, για να το πω έτσι, οι χώρες ε, ε, από τις δύο τελευταίες διευρύνσεις υπέγραψαν τη Συμφωνία για τη ε, ε, παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Η κυρία ε, Λάστραμ έχει το λόγο. Σνίμπερα Λάστραμ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Γέλεβα. Στην αρχή της σημερινής ακρόασης μιλήσατε για τις επιπτώσεις των θεομηνιών των περιβαλλοντικών καταστροφών, ιδιαίτερα στις φτωχές χώρες. Και είπατε ότι θέλετε ε, να δημιουργήσετε μεγάλες ε, δυνατότητες με συντονισμό που είναι λέτε ακρογωνιαίος λίθος. Τι σημαίνουν όλα αυτά παρακαλώ συγκεκριμένα, μπορείτε να μας εξηγήσετε. Έχετε το λόγο κύριε Αγέλα. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας και θα σας έλεγα ότι ο συντονισμός πραγματικά είναι ε, η λέξη κλειδί εδώ. Mm. Όχι μόνο επειδή Θέλω να συνδυάσω αυτά τα τρία στοιχεία στο χαρτοφυλάκιό μου που εντάσσονται πλέον και τα τρία, αλλά διότι οι κρίσεις έχουν γίνει πλέον τόσο περίπλοκες, ώστε να χρειάζεται πραγματικά πολύ μεγάλο συντονισμός με τους επιτόπου ε, επιρογνώμονες, ειδικού ανθρώπους που ζουν εκεί. Και είναι πολύ σημαντικό όντως τα θέματα αυτά να τα συζητούν όχι μόνο το κέντρο, εδώ οι υπηρεσίες μας και είναι καλά προετοιμασμένες για τα διάφορα ε, θέματα, τις διάφορες θεομηνίες και την απόκριση που πρέπει να δίνεται στην εκάστοτε κρίση, αλλά να έχουμε και συγκεκριμένη συνεργασία, όχι μόνο σενάρια για τις ε, ξεχασμένες κρίσεις ή για τις παγκόσμιες κρίσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε τελική ανάλυση να γνωρίζουμε και τι λένε οι άνθρωποι εκεί και να υπάρχει πολύ καλός συντονισμός. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι καταρχάς έχουμε πάρα πολύ καλές υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλό επαγγελματισμό. Αλλά έχουμε και εκατοντάδες εμπειρογνωμόνων επί τόπου που σε κάθε περίπτωση είναι σε θέση να κάνουν καλές αναλύσεις της εκάστοτε ε, κατάστασης για το ποια είναι οι αναγκαίες δράσεις και ποιοι είναι οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι. Σε λίγες μόνο ώρες μπορούν να τα αναλύσουν όλα αυτά. Έχετε συμπληρωματική ερώτηση, παρακαλώ, κυρία Σνίμπε. Όχι. Καλώς. Ε, ο, ο λόγος τώρα στην κυρία Τόγια, Πατρίσια. Sostituisco Τόγια, grazie. Ναι, εγώ λέγομαι Τόγια και αντικαθιστώ την άλλη κυρία. Κυρία Γέλεβα, απαντώντας στο Λιμισελ, Μισελ, παρεμπιπτόντος αναφερθήκατε στο θέμα της ασφάλειας των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις. Ένα ε, ερώτημα πολύ σαφές. Ξέρουμε ότι αυξάνονται οι επιθέσεις εναντίον της ζωής των εργαζομένων αυτών θεωρείται ότι εκφράζουν τις ε, δυτικές ας πούμε, πολιτικές. Κι όμως είναι αποφασιστική για τη διανομή της βοήθειας, για την ε, επιτόπια παρέμβαση. Θα ήθελα λοιπόν να μου απαντήσετε άμεσα τι σκοπεύετε να κάνετε εσείς, να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα της αύξησης των επιθέσεων εναντίον των εργαζομένων στις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Ε, αναφέρθηκα στην ασφάλεια των εργαζομένων αυτών, που είναι μία από τις προτεραιότητές μου. Και το 2008, πάνω από 100 άτομα σκοτώθηκαν. Και έχασαν τη ζωή τους με το χειρότερο τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ένα ασφαλές πλαίσιο μέσα στο οποίο θα δουλεύουν οι εργαζόμενοι αυτοί για τις επιχειρήσεις των οργανώσεων ανθρωπιστικής βοήθειας και είμαι έτοιμη να συνεργαστώ με όλους τους αρμόδιους φορείς στις εν λόγω χώρες. Είμαι έτοιμη να εξασφαλίσω καλό διάλογο με όλους τους ενδιαφερομένους φορείς μη κρατικούς ή κρατικούς φορείς στις χώρες αυτές. Γιατί βεβαίως γνωρίζω ότι οι σειράξει είναι επικίνδυνε. Και βεβαίω θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προετοιμάσουμε του εργαζόμενου αυτού. Την προηγούμενη εβδομάδα συναντήθηκα με εκπροσώπου των μη κυβερνητικών οργανώσεων και συζητήσαμε ανοιχτά. Ε, ανησυχούν πραγματικά γιατί συχνά είναι δύσκολο να βρουν ε, καλά στοιχεία εργαζόμενους με προσόντα. Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν σε ό,τι αφορά την κατάρτιση των ανθρώπων αυτών. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Κυρία Τρόια, έχετε, ε, τη έχετε και άλλη ερώτηση. Το, η ενδιάμεση έκθεση του 2010 του ΟΗΕ, τι σχέση θα σκοπεύετε να έχετε με τον ΟΗΕ, ε, τι ποια διάσταση σκοπεύετε να προωθήσετε με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι πολύ σημαντικό στοιχείο του δικτύου μας. Δουλεύουν επί τόπου, εκεί όπου υπάρχει το πρόβλημα. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν πραγματική εμπειρογνωμοσύνη, είναι προετοιμασμένες θα ενδυναμώσω την ε, συνεργασία μαζί τους. Υπάρχουν οι διαδικασίες, υπάρχουν οι κανόνες για την επιλογή των ε, ατόμων που θα εργαστούν σε αυτές. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος που εκπροσωπείται από την κυρία Στρέλα. Κυρία το 2006 το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα για τις θεομηνίες. Ψήφισμα στο οποίο ζητούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, καταθέσει οδηγία για την προστασία και την πρόληψη των δασοπυρκαγιών και μάλιστα γινόταν λόγος για ευρωπαϊκό παρατηρητήριο για ε, την παρακολούθηση των πυρκαγιών, της ξηρασίας και των πλημμυρών προτίθεστε να καταθέσετε μια τέτοια οδηγία για να χαρτογραφηθούν οι περιοχές και να εντοπιστούν οι περιοχές ακριβώς που κινδυνεύουν. Και επίσης θέλω να γνωρίζω τι φρονείτε για τη δημιουργία αυτού του παρατηρητηρίου. Παρακαλώ, κυρία Γέλεβα. Αυτό το κέντρο πληροφόρηση είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την πολιτική προστασία και τον αντίστοιχο μηχανισμό στην Ένωση και όντως θα πρέπει να ενισχυθεί. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι το Κοινοβούλιο υποστηρίζει αυτές τις προσπάθειες, το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και ε, άλλα πολιτικά έγγραφα το υποστηρίζουν. Και με τη συνδίκη της Λισαβόνας έχουμε και τη ρήτρα αλληλεγγύης, καθώς επίσης και τη δυνατότητα να ενισχύσουμε το μηχανισμό αυτό. Για την αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών αλλά και εκτός της Ένωσης. Συγκεκριμένα έρχομαι στην ερώτησή σας. Βεβαίως, είμαι πρόθυμη, αν είναι αυτή η επιθυμία του Κοινοβουλίου, ακούγοντας προτάσεις σας και τις υποδείξεις σας, να καταθέσω σε καλή συνεργασία και με ανταλλαγή απόψεων ε, μια πρόταση και να επανέλθουμε την πρόταση αυτή ενώπιόν σας. Ναι, παρακαλώ, έχετε το λόγο κυρία Στρέλα. Ευχαριστώ πολύ. Μα ήταν πολύ συγκεκριμένη η ερώτησή μου. Κοιτάξτε, τι ρώτησα εγώ. Θα καταθέσετε σχέδιο οδηγίας για τη διαχείριση και την πρόληψη των πυρκαγιών. Υπάρχει αντίστοιχη οδηγία για θέματα πλημμυρών, για παράδειγμα. Um, Η οδηγία είναι πολύ βαριά νομοθετική πράξη. Βεβαίως υπάρχει ανάγκη να το συζητήσουμε και στο κολέγιο των επιτρόπων για να ε, κάνουμε πρόταση τέτοιου είδους στο Κοινοβούλιο. Εγώ θα ήθελα να ακούσω τις δικές σας προτάσεις ως Κοινοβούλιο, διότι γνωρίζω ότι το Κοινοβούλιο έχει προχωρήσει πολύ και έχει αναλάβει σημαντικέ πρωτοβουλίε για την ανακούφιση πληθυσμών που αντιμετωπίζουν έκτακτε καταστάσει. Αν είναι λοιπόν αυτή η επιθυμία του Κοινοβουλίου, θα τη μελετήσω πάρα πολύ προσεκτικά. Και τώρα... Τώρα οφθαλμοθυρία, catch the eye. Πεντάλεπτη. Με θέμα την μείωση του ανθρωπιστικού χώρου και την αύξηση του χώρου δικαίου, ανθρωπιστικού δικαίου. Μπέρμαν. 15 με 20 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επειδή υπάρχουν πολλές καταχρήσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πρώην Κονγκό, πώς αναλύεται το σφάλμα που συνέβη εκεί, τι φταίει. Ο στρατός του Κονγκό αποτέλεσε τελικά εγκληματικό όπλο ο ίδιος. Ποιο ευθύνεται για τα τρομακτικά αυτά λάθη. Κυρία Γελέβα, η κατάσταση στην Γάζα από ανθρωπιστική σκοπιά είναι εντυπωσιακή από κακή πλευρά 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι υποφέρουν και το κράτος του Ισραήλ δεν ε, επιτρέπει τη δίωδο της ανθρωπιστικής βοήθειας. Τι θα κάνετε εσείς με τους συναδέλφους σας για να πηγαίνει καθημερινά η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Ο κύριος Νιούτον Ντάν. Εδώ είμαι, κυρία υποψηφία. Οι κρίσει εξορισμού είναι ευνίδιε. και θα έχετε 27 κυβερνήσεις που δεν θα θέλουν να σας δώσουν χρήματα γιατί αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Εσείς πώ θα του αντιμετωπίσετε του 27 αυτού ή όσοι είναι που δεν θα σας πιστεύουν σε αυτά που τους λέτε ευνίδιω. Κυρία Αγία Λεβά, έχετε το λόγο για να απαντήσετε σε αυτές τις τρει ερωτήσει. Thank First Το πρώτο, το Κονγκό. Γνωρίζουμε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια υφίσταται πιέσεις, ε, περιορίζεται και θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε σε όλα τα επίπεδα και να προσπαθήσουμε να εντείνουμε, να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με τους ντόπιου ε, φορείς και θα είναι από τα πρώτα μου μελήματα σε περίπτωση που ε, εγκριθεί ο διορισμός από το Κοινοβούλιο. Για τη Λωρίδα της Γάζας θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι θα μεταβώ στη Λωρίδα της Γάζας και θα είναι από τις πρώτες μου επισκέψεις και πάλι αν επιβεβαιωθεί ο διορισμός μου, διότι ανησυχώ πάρα πολύ για την κατάσταση. Ε, Γνωρίζω ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα, ο αποκλεισμό, ας πούμε, αλλά και ε, η μη ε, άφηξη της βοήθειας εκεί. Το 95% του πληθυσμού εξαρτάται από τη δική μας ανθρωπιστική βοήθεια. Θα πρέπει να είμαστε πιο ενεργοί ε, σε προληπτικό επίπεδο και θα κάνω ό,τι μπορώ και θα πάω και η ίδια σας είπα στη Γάζα για να διαπιστώσω ιδίες όμαση. 27 κράτη-μέλη, είπατε, Ξέρω ως υπουργό Εξωτερικών της ε, Βουλγαρίας πόσο δύσκολο είναι να εργάζεται κανείς στο Συμβούλιο και να επιτυχάνει τη συνένεση. Πάντα υπάρχει μια ομάδα κρατών που δεν θέλουν να συμμετέχουν, δεν θέλουν να είναι γραμής γραμμή της πλειοψηφίας. Ε, νομίζω ότι είμαι καλή στον απίθο και έχω και την προθυμία ο κύριο Χάουιτ έχει το λόγο. Έχουν ζητήσει και άλλοι το λόγο, δύο. Ω υπουργό Εξωτερικών, πώς προωθείτε το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες και τι έχετε διδαχθεί από ε, αυτή σας την εμπειρία για τη μελλοντική ανθρωπιστική βοήθεια. Η κυρία Κέλλε. Ο κύριος Κέλλη, όχι η κυρία Κέλλερ. Καταρχάς, ε, συγχαρητήρια κυρία Γέλεβα, γιατί αντιμετωπίζετε δύσκολη κατάσταση και εσείς εδώ. Σας ερωτώ, πώς αποφασίζετε να δοθεί ανθρωπιστική βοήθεια σε χώρες όπως η Ζιμπάμπουε, για παράδειγμα, που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και κλπ. Η κυρία Στριφλέρ, παρακαλώ. Ναι, σε σχέση με αυτά που υπόθηκαν προηγουμένως για τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Λέτε ότι είναι προτεραιότητα. Κάθε μέρα βιάζονται 100 γυναίκες. Και μας λέτε ότι θα πάτε εκεί. Εγώ θέλω πιο συγκεκριμένες απαντήσεις. Το έχετε σκεφτεί, έχετε μας δώσετε ένα παράδειγμα για το τι θα μπορούσατε να κάνετε απέναντι σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Έχετε το λόγο για να απαντήσετε στις τρεις αυτές τις Uh, uh, Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πάρα πολύ σημαντικά σε όλες τις πολιτικές μας συζητήσεις. Ε, σας διαβεβαιώ ότι έχουμε πάρα πολλά θέματα που μας ε, απασχολούν ε, σε διάφορες κρίσεις, στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Ευρώπη, αλλά και εκτός της Ευρώπης. Έχω συμμετάσχει με τρόπο πάρα πολύ ενεργό ως υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Τώρα, για τις καταχρήσεις και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ζιμπάμπουε. Ε, ή σε άλλες περιοχές. Ε, βεβαίως πολλά μπορούμε να κάνουμε. Όπως σας είπα προηγουμένως, μπορούμε να αρχίσουμε από την άσκηση υγιούς διπλωματίας. για να ε, μας επιτρέψουν την πρόσβαση καν ε, στις ανθρωπιστικές μας οργανώσεις για ανθρωπιστική βοήθεια. Από εκεί και πέρα μπορούμε να προχωρήσουμε στην άσκηση πολιτικής πίεσης ε, στις αρχές των κρατών αυτών. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση για την κατάσταση των γυναικών στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό και τη σεξουαλική κακοποίηση ως γυναίκα πραγματικά πρέπει να σας πω ότι το θέμα ενδιαφέρει πάρα πολύ και θα δραστηριοποιηθώ έντονα σε αυτό, διότι ακριβώς δεν μπορούμε να επιτρέπουμε στον 21ο αιώνα τη χρυσή τέτοια βίας που να ασύζει στο φύλλο και σεξουαλικής κατοκοπής όπως είναι ο βιασμός ε, σε καιρούς πολέμου. Ε, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τέτοια φαινόμενα και θα καλέσω τις υπηρεσίες μου σε επίπεδο επιχειρησιακό να είναι πιο δραστήριες στην προστασία των γυναικών. Θα πρέπει να συνεχίσουμε, λέει, πρόεδρος και διακόπτη την ομιλήτρια. Ο κύριος Ιβο Βάιγκελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Είναι δύσκολο πράγμα να απαντάει κανείς συνεχώς και σε μία τόσο λίγο εμπνευστική ατμόσφαιρα σε ερωτήσεις. Αλλά νομίζω ότι ο πρόεδρος Μπαρόσο πρέπει να σας κάνει μία λεπτομερή, να ζητήσετε από τον πρόεδρο Μπαρόσο γνωμάτευση νομική για τις κατηγορίες που ακούστηκαν εναντίον σας. Τώρα άλλο θέμα, το Σουδάν και το Ισραήλ. Ήσασταν υπουργό Εξωτερικών, είστε έμπειροι πολιτικός, λοιπόν τι μπορείτε να κάνετε για να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα που δημιουργούν ή αντιμετωπίζουν οι δύο αυτές κυβερνήσεις. Ορίστε κυρία Γελέβα. Το ανθρωπι... Η ανθρωπιστική βοήθεια είναι ανεξάρτητη. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ζητούμε πρόσβαση για να μας δοθεί η δυνατότητα να χορηγήσουμε βοήθεια. Στην περίπτωση του Σουδάν ξέρω πολύ καλά ότι εκεί είμαστε πολύ δραστηροί εδώ και πολλά χρόνια η κατάσταση εκεί συνεχίζει να είναι κρίσιμη αν και αλλάζουν οι περιοχές όπου υπάρχει, μειώνονται οι παραβιάσεις αλλά Φυσικά δεν είμαστε ικανοποιημένοι γενικά, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο. Από τη δική μου πλευρά υπάρχει πάντα η διάθεση να πάμε επί τόπου, να δούμε, να συναντήσουμε τις πολιτικές αρχές εκεί. Για το Ισραήλ, σας είπα ήδη κάτι για τη Γάζα προηγουμένως. Και εκεί βλέπω πολλές δυνατότητες για να δραστηριοποιηθούμε, ακόμη και σε τεχνικό επίπεδο μιλώντας, σε συνεννόηση με όλους τους παράγοντες εκεί και ενδιαφερόμενους. Θα επισκεφθώ και τη Γάζα, αν διοριστώ. Και τη Γάζα. Τη λουρίδα της Γάζης. Η κυρία Θεό Καράους. Θεοχάρους. Θεοχάρους. Ευχαριστώ κυρία Γέλεβα. Είναι γνωστό ότι το AIDS είναι ασθένεια των φτωχών, αλλά επίσης είναι γνωστό ότι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας δίνει αντιϊκά φάρμακα δωρεάν σε ε, ασθενείς μόνο εφόσον υπάρχουν εργαστηριακές αναλύσεις και αιματολογικές. Αλλά τεράστιο ε, ποσοστό πληθυσμό θερούνται αυτή τη ιατρική υπηρεσία λόγω διαχείριση ανθρωπιστική βοήθειας και διαφθοράς. Αυτό το παράδειγμα δείχνει ότι είναι ε, κρίσιμο και αποφασιστική σημασία να ε, ξεπεράσουμε τη διαφθορά σε υψηλό επίπεδο και να πηγαίνει στις κοινότητες επιτόπου η ανθρωπιστική βοήθεια. Έχετε έναν τρόπο και την πρόθεση αυτά να τα κάνετε πράξη. Έχετε το λόγο, κυρία Γέλεβα. Η παροχή ιατρικής ε, φροντίδας είναι σημαντικό στοιχείο της συνεργασίας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η ανθρωπιστική βοήθεια ε, βασίζεται πάντα σε συγκεκριμένες ανάγκες και καθοδηγείται από αυτές. Και όταν υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες σε κάποιες χώρες, αναφερθήκατε στο AIDS, βεβαίως και θα δώσουμε τα απαραίτητα φάρμακα και την απαραίτητη φροντίδα υγείας. Η διαφθορά σε υψηλό επίπεδο είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και θα πρέπει να τη γνωρίζουμε. Αυτό δεν είναι δική μας υπόθεση να ξεπεράσουμε τη διαφθορά, αλλά μπορούμε να συνεισφέρουμε σε συνεργασία και να βεβαιωθούμε ότι τα φάρμακα που στέλνουμε εκεί και οι διάφορες υπηρεσίες να παρέχονται πραγματικά σε εκείνους που τα έχουν ανάγκη. Have the floor for um, Κυρία Θεοχάρου, εσείς έχετε την πρόθεση να συστήσετε μια ευρωπαϊκή ανθρωπιστική ομάδα κρούσης, task force, για να καλυφθούν όλες αυτές οι ανάγκες όταν χρειάζεται αυτό. Και στις ανθρωπιστικές κρίσεις. Ευχαριστώ. Σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας, ξέρετε ότι υπάρχει η ε, εθελοντική υπηρεσία, ανθρωπιστική, είναι επιπλέον ε, έργο. Τώρα, για την επιπλέον ομάδα κρούσης, Task Force για ε, τη φροντίδα υγείας, είναι καλή πρωτοβουλία, να τη σκεφτούμε, πολύ χρήσιμη ενδεχομένω, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε και να είμαστε και ρεαλιστές γιατί δεν έχουμε πόρους επιπλέον για αυτή την προσπάθεια. Parole est maintenant à Madame, à Monsieur David Maria Σασόλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, δεν είμαι πολύ ικανοποιημένο από τι απαντήσει σα για την ασφάλεια των εργαζομένων σε πολλές περιοχές ε, όπου δραστηριοποιούμαστε μέσω διαφορών οργανώσεων. Τι θα προτείνετε στην ύπατη ε, επίτροπο και στον Επίτροπο Ανάπτυξης για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα. Κυρία Γέλεβα, έχετε το λόγο. Όπως είπα ήδη, θα πρέπει να δουλέψουμε σε δύο επίπεδα ασφάλεια για τους εργαζομένους, να βελτιώσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο εργάζονται και χρήσιμο θα ήταν για να γίνει κάτι τέτοιο, να έχουν καλύτερη εκπαίδευση, κατάρτιση, ασκήσεις και εδώ, στο αρχηγείο μας, ας πούμε, εντός αγωγικών, αλλά και επιτόπου στις διάφορες χώρες. Επίσης, θα πρέπει να ζητήσουμε από τις ε, τρίτες χώρες να σεβαστούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Γιατί αυτό είναι το πλαίσιο, αυτό είναι το δίκαιο που μας επιτρέπει να δώσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια, να την παραδώσουμε. Αυτά τα δύο επίπεδα θα πρέπει λοιπόν να συνδυαστούν. Αναφερθήκατε στην Αντιπρόεδρο και είπατε εκπρόσωπο την κυρία Άστον Ελπίζω εν καιρό να έχουμε καλή συνεργασία και, για τα θέματα του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου. Κύριε Σασόλη, έχετε συμπληρωματική ερώτηση. Στο Νότο, στο Σουδάν, συγγνώμη, Υπάρχει ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά λιγότερο το 50% του πληθυσμού έχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Τι σκοπεύετε να κάνετε, ούτω ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση α, να μην δίνει απλώ κονδύλια, αλλά να παίξει ένα ρόλο κλειδί για να βελτιωθεί η κατάσταση εκεί, στο Σουδάν. Κυρία Γέλεβα. Το Σουδάν αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες προβλήματα με τους πρόσφυγες, ε, με τους εσωτερικά εκτοπισμένους, προβλήματα με το πόσιμο νερό, με την ε, παροχή σύντησης. Και η Κομισιόν ξέρετε πολύ καλά ότι χρηματοδοτεί επιχειρήσεις, επιτόπου, εδώ και πολλά χρόνια. Γνωρίζουμε ποια είναι τα προβλήματα στο Σουδάν και το Σουδάν ε, συμπεριλαμβάνεται στο ετήσιο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζουμε την κατάσταση και παρόλα αυτά θέλουμε να δώσουμε με σωστό τρόπο βοήθεια. Ε, θέλουμε να εξασφαλίσουμε βέβαια και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ την κυρία Γέλεβα για το διορισμό της, για μια δουλειά που προωθεί τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συχνά μιλάμε για αυτές τις αξίες εδώ, σε αυτό το χώρο, σε αυτό τον οίκο. Είπατε κάτι προηγουμένως στο οποίο θέλω να επανέλθω. Είπατε ότι θέλετε να καταπολεμήσετε τη σεξουαλική βία που έχει γίνει όπλο, όπως είπατε. Θα ήθελα σας παρακαλώ να πείτε λίγα λόγια παραπάνω για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Κυρία Γέλεβα, έχετε το λόγο. Για τα θύματα σεξουαλικής βίας και για τη βία εναντίον συγκεκριμένου φύλου έχουμε συγκεκριμένα μέτρα. Ειδικά καταφύγια πούμε, για γυναίκες και κορίτσια που έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής βίας. Επίσης, ε, προβλέπουμε ε, ψυχολογική υποστήριξη, βοήθεια σε επίπεδο υγείας ανάλογα με τα συγκεκριμένα προβλήματα αναπερίπτωση. Αυτό ακριβώς κάνουμε στο Κονγκό. Και σε πολιτικό επίπεδο σκοπεύω να δώσω στο Κοινοβούλιο ένα κείμενο πολιτικής για τις ε, τομεακές πολιτικές που μπορούν να αφυπνίσουν τον κόσμο για αυτές τις ε, σεξουαλικές τα σεξουαλικά βασανιστήρια, τη σεξουαλική βία και για το γεγονός ότι η σεξουαλική βία χρησιμοποιείται ως όπλο σε διάφορες σειράξεις. Επίσης υπάρχει υπάρχουν και καλές πρακτικές για το πώς θα δώσουμε βοήθεια στα θύματα. Έχετε δεύτερη συμπληρωματική ερώτηση? Όχι. Ο κύριος Νόισερ. Κυρία Γέλεβα, στη νέα, στο νέο πρόγραμμα δράσης Αφγανιστάν-Πακιστάν της Ένωσης του περασμένου έτους της Άνοιξης ε, γίνεται λόγος για τη βοήθεια προς την αυτοβοήθεια. Ε, συγκεκριμένα αυτό τι σημαίνει για το Αφγανιστάν. Ε, τα μέτρα του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων και της Ένωσης πώς θα τα συντονίσετε. Και δεύτερη ερώτηση, τι θέλετε να κάνετε συγκεκριμένα έτσι ώστε να προστατεύονται και να ενισχύονται περισσότερο και να προβάλλονται περισσότερο οι πολιτικές μας δράσεις που είναι και πάρα πολλέ στο Αφγανιστάν απέναντι στι στρατιωτικές. Ε, έχετε το λόγο. Το Αφγανιστάν είναι πραγματικά μια χώρα που μας απασχολεί πάρα πολύ και δίνουμε και πάρα πολλά χρήματα. Η βοήθεια στην αυτοβοήθεια είναι πολύ σημαντική και πρέπει να σας πω ότι ακριβώς στο Αφγανιστάν έχουμε ένα μείγμα ανθρωπιστικής βοήθειας και στρατιωτικής δράσης και ως έτσι θα πρέπει να το βλέπουμε και αυτό, αυτό μας απασχολεί όμως γιατί γίνεται μια σύγχυση ανάμεσα στην ανθρωπιστική μας παρουσιακή και στη στρατιωτική. Ε, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, να πούμε ποια είναι η πολιτική μας δράση οι μη στρατιωτικοί δηλαδή και πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερο συντονισμό με τους στρατιωτικούς. Για να έχουμε δράση ανθρωπιστική και να βοηθούμε τις κοινότητες θα πρέπει να έχουν και πρόσβαση οι άνθρωποι αυτοί. Αλλά να μην θεωρούν ως δική τους δουλειά οι στρατιωτικοί να παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια. Απλώς και μόνο να εξασφαλίζουν την πρόσβαση. Αλλιώς αντιτίθεται αυτό ε, στις βασικές μας ε, αρχές. Είναι πολύ σημαντικό για τη διεθνή κοινότητα να έχουμε και πολιτική δράση εκεί, ε, χέρι με χέρι με τη στρατιωτική χωρίς να συγχέονται αυτά τα δύο, επαναλαμβάνω. Και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και είμαι πρόθυμη να βοηθήσω προς την κατεύθυνση αυτή για να προωθήσουμε την ανθρωπιστική μας ε, δράση και την παροχή βοήθειας προς τις επιτόπου κοινότητες. Σύντομη συμπροματική ερώτηση. Στην ανθρωπιστική βοήθεια λοιπόν και σε αυτά που θέλει τώρα η κυβέρνηση Καρζάη, τη ε, διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης. Θα θεωρούσατε σκόπιμο να προσεγγίσουμε με τριοπαθείς τα Λιμπάν και να αρχίσουμε ένα διάλογο μαζί τους. Έχετε το λόγο. Εξ όσων γνωρίζουμε, οι Ταλιμπάν ελέγχουν το 60% του συνόλου της επικράτειας της χώρας για την ανθρωπιστική δράση είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πρόσβαση ε, στα εδάφη αυτά και να υπάρχει και ασφάλεια για την ανθρωπιστική βοήθεια και την παροχή της. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν σε τεχνικό επίπεδο είμαστε υποχρεωμένοι να συνεργαζόμαστε με όλους τους ε, φορείς. Αν αυτό είναι χρήσιμο και ε, βοηθάει και βελτιώνει και τη ζωή ε, και εξασφαλίζει την ακαιρεότητα των ε, ανθρώπων που εργάζονται στις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Κυρία Στριφλέρ. Στην επιστολή του κυρίου Μπαρόζο προκύπτει ότι ο συντονισμός για την πολιτική προστασία ε, τη χάν διαχείριση από την ΕΚΟ. Αυτό σημαίνει ότι ένα τμήμα των ε, επιχειρήσεων ε, θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν κάποια στιγμή από τον προπολογισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας ε, και ποια είναι η θέση σα. Μικρόφωνο. Έχουμε πολύ σαφείς γραμμές στον προπολογισμό. Έχουμε την ανθρωπιστική βοήθεια, με ένα προπολογισμό 700 εκατομμύρια ευρώ και η πολιτική προστασία έχει έναν άλλο προπολογισμό. Δεν υπάρχει πρόβλημα για συγχώνευση. Μπορούμε να έχουμε περισσότερο συντονισμό τώρα ανάμεσα στα δύο επίπεδα. Και μπορούμε να έχουμε να δίνουμε ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτική προστασία με συμπληρωματικό τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Αλλά δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε και τους δύο προϋπολογισμούς ε, για το ίδιο πράγμα. Η φύση των δύο γραμμών προϋπολογισμού είναι τελείως ε, διαφορετική. Κυρία Στίφλερ, έχετε συμπληρωματική ερώτηση. Όχι. Θα περάσουμε τώρα στην ακρόαση ε, συμμετέχει τώρα η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ε, εκπροσωπείται από την κυρία Χάουταλα. Η ασφάλεια των ανθρωπιστικών οργανώσεων και των εργαζομένων τους ε, συζητήθηκε ήδη. Κυρία Γέλεβα, πώς θα εξασφαλίσω μεγαλύτερη προστασία σε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα ε, πολυάριθμων ανθρώπων που ζουν σε στρατόπεδα γιατί είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι. Τι πρόγραμμα έχετε για να εξασφαλίσουμε τα βασικά θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά τους. Ε, θεωρείτε ότι η κατάρτιση, η συστηματική κατάρτιση των ε, ανθρώπων που δουλεύουν ε, σε αυτά τα στρατόπεδα είναι τμήμα αυτής της προσπάθειας, κυρία Γέλεβα. Απαντήστε. η κατάρτιση μέσα στα στρατόπεδα για τους ε, εσωτερικά εκτοπισμένους πληθυσμούς είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο. Τα άτομα αυτά συχνά ζουν για μεγάλες περιόδους ε, στα στρατόπεδα. Δεν θα πρέπει να τα πιέζουμε λοιπόν. να επαναπατριστούν ε, στην περιοχή από την οποία προέρχονται, στη χώρα από την οποία προέρχονται. Θα πρέπει ο επαναπατρισμός να γίνεται εθελοντικά. Θα πρέπει να παρέχουμε κατάρτιση, ε, μαθήματα για να τους διδάξουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για το τι μπορούν να διεκδικήσουν. Κυρία Χάουταλα, έχετε δεύτερη συμπληρωματική ερώτηση. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε, ναι. Το να εγγυηθούμε τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση. Έχετε κάποιες ιδέες για το πώς θα εξασφαλίσουμε αυτά τα δικαιώματα. Διάβασα και προετοιμάστηκα για αυτή την ακρόαση, το μάτι μου έπεσε σε μια σημαντική φράση. Ότι οι γυναίκες σε αυτές τις χώρες, σε χώρες όπου υπάρχουν σειράξεις, αυτές είναι οι φορείς της αλλαγής. Όταν υπάρχει βία εναντίον γυναικών και κοριτσιών, θα πρέπει εμείς να δραστηριοποιηθούμε, να διδάξουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, αυτές τις γυναίκες και τα κορίτσια, τα δικαιώματά τους. Να τις βοηθήσουμε κοινωνικά και ψυχολογικά. Είναι πολύ δύσκολο να μιλήσουμε στα θύματα σεξουαλικής βίας. Είναι πολύ δύσκολο να επανενταχθούν στην πραγματική ζωή να συνδεθούν με την προηγούμενη ζωή τους. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να τις βοηθήσουμε και να τις υποστηρίξουμε. Και τώρα φτάνουμε στο follow-up και στις ερωτήσεις τις ε, συμπληρωματικέ τρίτο και τέταρτο γύρο σε σχέση με ερωτήσεις που έχουν τεθεί προηγουμένως. Έχουμε εννέα λεπτά, αλλά δεν έχω λάβει γραπτές ερωτήσεις. Έχετε 30 δευτερόλεπτα για να μου τις ε, στείλετε. Voilà, je laisse quelques secondes. Et si il n'y a pas de follow-up question... Αν δεν υπάρξουν τέτοιες ερωτήσεις follow-up, θα συνεχίσουμε με το τελευταίο γύρο ερωτήσεων. Monsieur Berman, s'il n'y a que vous, je pense que vous pouvez la poser directement vous-même. Thank you, Madam Ο κύριος Μπέρμαν. Κυρία Ζέλεβα, θα ήθελα πραγματικά να σας παρακαλέσω να είστε πιο συγκεκριμένοι στην ανάλυση σας. Τι πήγε στραβά με την υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών στη δράση του στρατού του Κονγκό. Τεράστια ε, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν τελείως ανεπαρκής η υποστήριξη από τον ΟΗΕ. Τι πήγε στραβά, παρακαλώ συγκεκριμένα πείτε μας πώς δεν θα ξαναγίνει αυτό στο μέλλον. Έχετε το λόγο κυρία Σάλεβα. So, I'm here really not uh, to, Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω βάλει υποψηφιότητα για τη θέση του Γενικού Διευθυντού των Υπηρεσιών μας. Και πιστέψτε με ότι δεν γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες στη ε, συγκεκριμένη αυτή περίπτωση. Αλλά είμαι πρόθυμη να σας διαβεβαίωσω ότι θα επανέλθω με συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Bon, nous commençons maintenant la dernière euh, ronde. Λοιπόν, περνούμε στο τελευταίο γύρο ερωτήσεων και το λόγο έχει ο κύριος Γκερέρο. Ευχαριστώ. Κυρία Ζέλεβα, η ασφάλεια των εργαζομένων στην ανθρωπιστική βοήθεια είναι όλο και πιο κρίσιμη για την ίδια την αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Είπατε ότι πέρυσι έχασαν τη ζωή τους πάνω από 100 εργαζόμενοι, περισσότεροι από κοιονόκρανους τότε. Και πρόσφατα έχουν απαχθεί πολύ σε διάφορα μέρη του κόσμου, σε διάφορα κράτη όπου ε, ασκούν αυτή την ανθρωπιστική τους δράση. Και χρειάζονται λοιπόν οι άνθρωποι αυτή η ευρωπαϊκή προστασία και προστασία της Ένωσης. Γι' αυτό σας ερωτώ, ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που θα υλοποιήσετε για να αυξηθεί αυτή η προστασία και αν συμπεριληφθεί αυτό στο σώμα των Ευρωπαίων εθελοντών. Έχετε το λόγο κύριε Ζέλεβα. Σε ό,τι αφορά ε, το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών είναι πάρα πολύ σημαντικό όντως και θα πρέπει να κάνουμε πολύ προσεκτική ε, πρόταση μετά από μελέτη. Θα πρέπει να αποφύγουμε λοιπόν να στέλνουμε σε επικίνδυνες καταστάσεις εθελοντές, σε πόλεμες σειράξεις. Ε, θα Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα η ασφάλειά τους ε, των εργαζομένων στις ανθρωπιστικές μας ε, δράσεις. Και ως προς την προστασία τους θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο που έχουμε στη δράση μας. Και βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί σε πολιτικό επίπεδο να καταγγέλει ε, τις παραβιάσεις και το μη σεβασμό του ανθρωπιστικού δικαίου γιατί είναι προϋπόθεση καν για να ασκήσουμε σωστά επιτόπου την ανθρωπιστική μας δράση. Και είμαι πρόθυμη να εργαστώ πάρα πολύ στενά με τη Βαρονή ε, Άστον για να απευθυνθούμε σε ε, υψηλό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το σεβασμό του διεθνού ανθρωπιστικού δικαίου, του διεθνού ανθρωπιστικού χώρου, για να μπορούν να εργάζονται ε, με ασφάλεια, με μεγαλύτερη ασφάλεια οι άνθρωποι μα εκεί. Ο κύριος Γκερέρο, ναι. Κανένα χρονοδιάγραμμα έχετε υπόψη σας πότε περίπου θα συσταθεί το σώμα των Ευρωπαίων Εθελοντών. Madame vous avez Κυρία Ζέλεβα, έχετε το λόγο. Η συνθήκη της Λισαβόνας ορίζει ότι είναι πολύ ε, σημαντικό αυτό το έργο μας. Μας λέγω, διότι θα επανέλθω με πρόταση, το πιθανότερο, στην Επιτροπή σας και αναμένω η πρόταση να είναι έτοιμη πριν το 2011 που ε, γνωρίζετε ότι είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού. Θα ήθελα να μοιραστώ με το Κοινοβούλιο αυτή την εμπειρία και να ε, ανταλλάξω και απόψεις με την ε, αξιότιμη επιτροπή σας για τον τρόπο με τον οποίο αυτή η πολιτική ιδέα θα μεταφραστεί στην πράξη συγκεκριμένα. La parole est maintenant Η κυρία Στρίφλερ. Μάλιστα. Μας λέτε επανειλημμένα ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο είναι σημαντικό, ότι πρεσβεύεται το α, θα πατέ επί τόπου. Ε, αυτό είναι το φυσιολογικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφωνήσει για το ανθρωπιστικό δίκαιο από το 2005 ε, να φροντίζει να γίνεται σεβαστό το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Αυτές οι δεσμεύσεις ε, είναι γνωστές, είναι πάρα πολλές οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου και επιδεινώνεται η κατάσταση. Λοιπόν, συγκεκριμένα κυρία μου, συγκεκριμένα τι θα κάνετε για να σέβονται το ανθρωπιστικό δίκαιο. Με χρηματοδότηση, με... Ε, με ποιους, σε ποιους θα προσφύγετε, ε, θα κάνετε κανένα διαγωνισμό, πρόσκληση, εκδήλωση ενδιαφέροντος, σε ποιους θα απευθυνθείτε. Έχετε το λόγο. Θα μπορούσα να φανταστώ κατά τη διάρκεια του έτους ακόμα να οργανώσουμε ένα μεγάλο διεθνές φόρουμ για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Έχω συζητήσει την ιδέα αυτή με τον προκάτοχό μου, τον Λουί Μισελ, και νομίζω θα ήταν καλή ιδέα να καλέσουμε όλους τους ενδιαφερομένους φορείς. Άλλη δυνατότητα θα ήταν να προσπαθήσουμε να πείσουμε περισσότερο όλο και περισσότερο ε, οργανώσεις και ε, δημόσιες αρχές τρίτων χωρών, όλο και πιο πολλούς, ε, σε χώρες που δίνουμε βοήθεια ανθρωπιστική για να καταλάβουν, να συνειδητοποιήσουν ποιε είναι οι ανθρωπιστικές αρχές και πώς θα πρέπει να γίνεται σεβαστό το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Ταυτόχρονα θα ήθελα να θέσω αυτό το ζήτημα και στα πλαίσια του Συμβουλίου Υπουργών Αμήνης για να ε, ζητούν και τα κράτη-μέλη από τους εταίρους μας περισσότερο σεβασμό. Κυρία Στριφλέρ, έχετε συμπληρωματική ερώτηση. Όχι. Η κυρία Ντεκεζέρ. Επιτρέψτε μου, κυρία Υποψήφια Επίτροπε, να επανέλθω στο θέμα της γάσας. Οι απαντήσεις σας δεν με πείσανε. Τι είπατε επί της ουσίας. Είπα ότι θα πρέπει να είμαστε πιο δραστήριοι, ότι θα πάω επί τόπου, θα δουλέψω με τους τοπικούς φορείς. Αυτά έκανε και ο κύριος Μπιμισό και η κυρία Φέρερο Βάντνερ. Με πολύ καλό τρόπο μάλιστα. Ε, όταν ε, λέτε ότι θα γίνετε δραστήρια, ε, τι εννοείτε, ότι οι προκάτοχή σας δεν ήταν αρκετά δραστήρι. Ε, το θέμα δεν είναι ότι η ανθρωπιστική βοήθεια μπλοκάρεται στη Γάζα. Εγώ ήθελα να ακούσω από εσά μια ανάλυση για την κατάσταση. Σας παρακαλώ, πείτε μας δύο λόγια Κυρία Γέπεβα. Είναι γνωστό βεβαίως ότι εδώ και πολλά χρόνια η διεθνής ε, κοινότητα και πολλοί φορείς, μεταξύ των οποίων και οι επίτροποι, ο κ. Λουί και η κυρία Φρέρο Βάλτεν, προσπάθησαν να δραστηριοποιηθούν. Δεν, έκαναν τίποτα. Απλώς η κρίση είναι παρατεταμένη. Ο καθένας έκανε ό,τι μπορούσε για να βοηθήσει. Δεν μπορείτε να περιμένετε ότι η Κομισιόν ή εγώ ως Επίτροπος θα είμαστε σε θέση να επιλύσουμε τα πάντα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να δώσουμε ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή αυτή και αυτό είναι πρόβλημα. Αν καταφέρουμε να δώσουμε, να χορηγήσουμε ανθρωπιστική βοήθεια, αυτό θα ήταν πραγματική πνοή και ανάσα πνο... Ε, ζωής για τον πληθυσμό εκεί. Το 95% του πληθυσμού στη Γάζα εξαρτάται από τη βοήθειά μας. Γι' αυτό λοιπόν δίνουμε ρευστό για τη δουλειά που κάνει ο ντόπιο πληθυσμό. Για καθαρισμό των πόλεων, για την αποκομιδή των σκουπιδιών. Πολύ χρήσιμο είναι αυτό. Δεν μπορώ να σας πω ότι εγώ θα βρω τη λύση πανάκια. Κύριε Ντεκαϊζέρ, έχετε δεύτερη ερώτηση. με που δεν ακούω, κυρία Γέλεβα, να, μου λέτε, να λέτε τίποτα για τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσετε, για τα μέσα που θα χρησιμοποιήσετε για να ασκήσετε πίεση. Νομίζω ότι υπάρχουν τέτοια εργαλεία. Αυτό περίμενα να ακούσω από εσά. Και αυτό περίμενα να ακούσω όταν απαντήσατε στο ερώτημα του Λουί Ο κύριο Λουί Μισελ σας ρώτησε τι εργαλεία θα χρησιμοποιήσετε, τι σχέσει θα έχετε με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Κύριε Γελέβα. Ήδη χρησιμοποιούμε το εργαλείο σταθερότητας. Ε, χρησιμοποιούμε όλα τα κανάλια που έχουμε για τον πολιτικό διάλογο. Αλλά η κατάσταση είναι περίπλοκη. Σας είπα ήδη προηγουμένως ότι δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα λύσω το πρόβλημα. Κανένας δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να φτάσει η βοήθειά μας επί τόπου. και να μετριαστούν τα δεινά του τοπικού πληθυσμού. Υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία στη διάθεσή μας. Αλλά καταρχάς πρέπει να έχουμε πολιτική θέληση για να επιλύσουμε το πρόβλημα και αυτό το ξέρετε πολύ καλά και εσείς όπως και εγώ. Κύριος Κάσλερ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Ζελεβά. Παρά τις διεθνείς προσπάθειες, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίω κάθε άλλο παρά εθαρρυντική είναι. Παράδειγμα, η ελευθερία τύπου, η ελευθερία θρησκείας, η ελευθερία γνώμης σε κάποια κράτη-μέλη καταπατώνται. Πρόσφατο πρόβλημα και παράδειγμα το Ιράν. Εμείς καλούμαστε παντού στον κόσμο να βοηθήσουμε για την προστασία των ε, παγκοσμίων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και σας ερωτώ, εσείς πώς θα συνεισφέρετε, ποια είναι η προτεραιότητά σας στον τομέα αυτό. Ένα-δυο παραδείγματα μπορείτε να μας δώσετε στην ανθρωπιστική βοήθεια και επίσης να μας πείτε τι γίνεται ε, με τις κυρώσεις, αν υπάρχουν κάποιες κυρώσεις ή αν συνδέεται με την επιβολή κυρώσεων κάποια βοήθεια, η αιρεσιμότητα. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Έχουμε συμφωνίες με τρίτες χώρες που είναι σημαντικό εργαλείο για να ασκούμε και επιρροή προς την κατεύθυνση αυτή. Για την ασφάλεια των εργαζομένων στην ανθρωπιστική βοήθεια. Μας σας είπα τις προτεραιότητες στην αρχή της τοποθέτησής μου, ορισμένες προτεραιότητες έκκληση για μεγαλύτερο σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. για τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας Αυτό μπορεί να γίνει με εφαρμογή νέων μεθόδων. Σας είπα και προηγουμένως, αυτόν τον καιρό Είμαστε σε ένα πειραματισμό, αλλά έχουμε και πολύ καλή πρακτική με ε, τη χρήση νέων τεχνολογιών σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των εργαζομένων στην ανθρωπιστική βοήθεια σε ε, διάφορα κράτη. Για τον νέο εξοπλισμό, όλα αυτά μπορούμε να τα εφαρμόζουμε στην εργασία μας. Ε, μου λένε επίσης οι υπηρεσίες μου ότι έχουμε ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου, ηλεκτρονικού οικονομικού ελέγχου. Αυτό θα βελτιώσει ε, και την αποτελεσματικότητα της εργασίας μας. Κύριος Κάσλε, έχετε συμπραγματική ερώτηση. Το τελευταίο παράδειγμα θέλω να σας ρωτήσω. Στο λογιστικό έλεγχο ή στην καταπολέμηση των κρίσεων, τι ρόλο βλέπετε για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις ή τις μεγάλες ε, φιλανθρωπικές οργανώσεις. Πώς βλέπετε και τη συνεργασία. Ε, Κυρία Ζέλεβα, όπως γνωρίζετε, η ανθρωπιστική βοήθεια δεν χορηγείται από μας με άμεσο τρόπο. Έχουμε δίκτυα. Και στο δίκτυο αυτό ανήκουν και μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Είναι πάνω από 185 συγκεκριμένα οι οργανώσεις αυτές και δεν είναι... μόνο οργανισμοί που εργάζονται επί τόπου και βοηθούν τους πληθυσμούς, αλλά είναι και σημαντική πηγή για ιδέες. Δεν τις χρησιμοποιούμε μόνο λοιπόν για λόγους επιμελητίας. Αυτά που είπατε είναι και εναλλακτικέ προτάσεις στις δικές μας εκθέσεις, στις δικές μας ε, σκέψεις και ιδέες. Ο κύριος Μίτσελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η διεθνή συνεργασία ε, είναι και ένα από, ε, μία από τις επικεφαλίδες στα χαρτοφυλάκια ε, μια σύγχυση και μια δυσκολία γιατί τρεις επίτροποι ασχολείστε με αυτό το θέμα. Ο δικός σας ρόλος ποιος θα είναι για τη διεθνή συνεργασία εκεί. Like Θα ήθελα να διαβιβάσω τον κύριο Μίτσελ ότι δεν υπάρχει καμία σύγχυση, κανένα περιθώριο για σύγχυση. Επανειλημμένα έχουμε συναντηθεί κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, προετοιμάζοντας την ακρόση, σχεδόν κάθε μέρα το κλάστερ, το λεγόμενο των επιτρόπων που ασχολούνται με θέματα εξωτερικών σχέσεων και υπάρχει και σαφής επιμερισμός των ε, αρμοδιοτήτων, των ρόλων μας και των καθηκόντων και μπορούμε να σας διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει καλύτερο συντονισμός και περισσότερη συνοχή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και η δική μου ξεχωριστή αρμοδιότητα θα είναι να ενισχύσω τη συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο με περιφερειακούς οργανισμούς, ΑΣΕΑΝ, Μέρκοσουρ και άλλους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Humanitarian, uh, όταν μιλάμε λοιπόν για σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και αν αποτύχει η σιωπηρή διπλωματία θα πρέπει να προχωρήσουμε στις ε, περιφερειακές οργανώσεις για να μας βοηθήσουν. Uh, για να ε, μας βοηθήσουν λέγω στην παροχή της ανθρωπιστικής μας ε, βοήθειας. Και σε πολλές περιπτώσεις χρειάστηκε να ενισχύσουμε τις δυνατότητες ε, γειτονικών κρατών να επηρεάσουν την ελόγω χώρα για να μπορέσουμε να περάσουμε και να δώσουμε την ανθρωπιστική μας βοήθεια. Για πρόσβαση μιλώ επιτόπου. Nous sommes maintenant. Non, ne pas. C'est Λοιπόν, περνούμε στην τελευταία ενότητα συμπληρωματικών ερωτήσεων. Γραπτές θα έπρεπε να μας είχατε δώσει τις ερωτήσεις, δεν έχω λάβει. Σας αφήνω λίγα δευτερόλεπτα, αν θέλετε να κάνετε ερώτηση. Ε, συμπληρωματική στην κυρία Ζέλεβα. Όχι, κανείς. Ετί αυτή η περιπτώση ολοκληρώνεται η ακρόαση ε, ως προς τις ε, ερωταποκρίσεις και θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Ζέλεβα για να κάνει τα καταληκτικά της σχόλια. Πέντε λεπτά το πολύ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, θέλω να σας ευχαριστήσω για την ενδιαφέρουσα αυτή ανταλλαγή απόψεων. Χάρηκα ιδιαίτερα για τη συνομιλία μας και προσβλέπω σε νέα συνάντησή μας, εάν διοριστώ. Όπως είπα και πριν, ως πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχω εκλεγεί δύο φορές στη Βουλγαρία είναι λοιπόν προσωπικό μου ενδιαφέρον να δημιουργήσω έναν στενό και έντονο διάλογο μαζί σας. Ως πολιτικό πρόσωπο θεωρώ ότι ο διάλογος είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και όχι μόνο αυτός, όχι μόνο ο διάλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά ιδιαίτερος με τους Ευρωπαίους πολίτες. Ε, Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα περισσότερα παραπάνω για να φέρουμε τους πολίτες κοντύτερά μας. Είμαι πεπισμένη ότι το Κοινοβούλιο θα υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια ως προτεραιότητα. Σε αυτή τη βάση η συνθήκη της Λισαβόνας μπορούμε να πούμε ότι μας έδωσε τη δυνατότητα καλύτερης προστασίας και φροντίδας των πολιτών και όλων όσων τη χρειάζονται διεθνώς για την αντιμετώπιση κρίσεων πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή να πλησιάσουμε τους θεσμούς με τους πολίτες για να τους δείξουμε ότι τα ευρωπαϊκά όργανα και οι θεσμοί για εκείνους εργάζονται και τους επιτρέπουν να ζουν σε ένα κλίμα ειρήνης, ασφάλειας και εμπιστοσύνης προς το μέλλον. Οι πολίτες έδειξαν ότι υποστηρίζουν στεναρά την Ένωση και η στήριξη όμως αυτή την χορηγούν εφόσον η Ένωση πραγματικά τους δίνει κάτι. Ενδιαφέρονται για τη ζωή της Ένωσης και τους συμπολίτε τους. Και επίσης για την τύχη των ασθενέστερων και πτωχοτέρων. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να, του διορισμού μου δηλαδή, να μπορέσω να καταστήσω τους Ευρωπαίους υπερήφαντους για τις αξίες μας διότι με τη βοήθειά τους, με την υποστήριξή τους τα ευρωπαϊκά όργανα δίνουν νέα ελπίδα και νέα αξιοπρέπεια σε όσους τη χρειάζονται περισσότερο. Θέλω οι λαοί μας να μπορούν να πούν με τη δική μου, και με τη δική μου συμβολή έσβησαν οι πυρκαγιές αυτές πριν να καταστρέψουν ανθρώπινες ζωές ή όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό έξω από τη χώρα τους να είναι περήφανοι όταν βλέπουν την ευρωπαϊκή σημαία ή ένα ευρωπαϊκό πανό σε έργα αναστήλωσης χωριών που έχουν πληγεί από θεομηνίες. Έτσι μόνο θα μπορέσω να πω ότι εκπλήρωσα τα καθήκοντά μου και το καθήκον μου προς τους ε, Ευρωπαίους πολίτες. Να δείξω δηλαδή, αν έχω δείξει, ότι οι πολίτες ενδιαφέρονται για τη δράση μας, ξέρουν ότι σώζουμε ζωές και την αξιοπρέπειά τους και τους δημιουργούμε νέες ελπίδες. Και ότι οι πολίτες και οι θεσμοί της Ευρώπης δουλεύουν χέρι το, με το χέρι. Χέρι-χέρι μάλλον. Και είναι υπερήφανοι οι για τους δε. Προσβλέπω με μεγάλο ενδιαφέρον στη συνεργασία μαζί σας για να ε, πραγματοποιηθούν όλα αυτά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας και ευχαριστώ και την υποψήφια Επιτροπογιά για τις απαντήσεις της. Πριν κηρύξω το πέρα συνεδρίαση, θυμίζω ότι οι συντονιστές συνεδριάζουν για την αξιολόγηση της παρούσης ακροάσεως και κλεισμένων των θυρών στις 8 η ώρα στην αίθουσα ASP 1G2. Λήξη συνεδρίασης, καλό σας βράδυ σε όλους.